Morning everybody. Via... Uh, Καλημέρα σας. Ξεκινάμε την σε διάμαξη. Παρακαλώ να συμφωνήσετε πριν από τις προφορίες σήμερα να προβούμε σε μια μικρή διόρθωση για το πρόγραμμα Creative Europe. γιατί έτσι μόνο μπορεί να κατατεθεί για έγκριση από την Ολομέλεια. Να δεχθείτε την συζήτηση του θέματος αυτού λοιπόν στην ημερήσια σα παρακαλώ για να σας εξηγήσω στη συνέχεια τι σημαίνει αυτό το διορθωτικό, το Creative Europe. Έχει κανείς αντίρρηση, όχι, ευχαριστώ πολύ. Πρακτικά τη συνεδριάσεως στις 20-21 Ιανουαρίου, 6 Φεβρουαρίου, 12-13 Φεβρουαρίου. Τα έχετε στα έγγραφά σας και προτείνω όσοι ήθιστε να θεωρηθούν εγκεκριμένα εφόσον δεν, προβούν, εφόσον δεν διατυπωθούν ε, ενστάσεις κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. Διερμηνία έχουμε εκτός από τα βουλγαρικά, πορτογαλικά, μαλτέζικα, εστονικά και ε, λίγο πολύ αυτές τις γλώσσες, όλες οι άλλες καλύπτονται. Και πάω στο 3α. Η γραμματεία σας έχει ενημερώσει και γραπτός ότι έχει αποστείλει μία πρόταση για διορθωτικό του άρθρου 24.6 του κανονισμού Creative Europe. Μία πρόταση για ε, διόρθωση του σημείου που έχει εσφαλμένα διατυπωθεί ως παραπομπή στο άρθρο 132 του Δημοσιονομικού Κανονισμού, να το αντικαταστήσουμε με μια παραπομπή στο άρθρο 131 του Δημοσιονομικού Κανονισμού. Αυτό είναι το διορθωτικό, γιατί ο Στίβεν πιστεύει ότι εμείς έχουμε τη σωστή παραπομπή από την Επιτροπή. Οι νομικοί έχουν εισαγάγει το εσφαλμένο άρθρο ως παραπομπή, Πρέπει λοιπόν να βρουν το θάρρος να χωρίσουν το σφάλμα τους και να κάνουν τη την διόρθωση. Το άρθρο 130 λέει ε, λέγεται από τη γραμματεία ότι δεν θα μπορούσε αν δεν γίνει η σχετική διόρθωση να καλύψει το Creative Europe. Συμφωνείτε λοιπόν να γίνει η διόρθωση για την, υπαγωγή για την παραπομπή στο 131, ούτως ή άλλως εμείς είχαμε δίκιο και πάλι μας αναγνωρίζετε λοιπόν και διορθώνεται το ε, άρθρο αυτό με την αναφορά, με την παραπομπή στο 131 του δημοσιονομικού κανονισμού, ώστε να μπορέσει να προχωρήσει και να λειτουργήσει το Creative Europe. Και πάμε στο σημείο 4 της τη διάταξη, τις νέες τεχνολογίες και ανοιχτή εκπαιδευτική πόρη. Καταλήν Σόρεν Ήβαν, εισηγητή. Η μόνη ψηφοφορία που έχουμε για σήμερα. Τον παρακαλώ Εάν θέλει να προσθέσει κάτι ο κύριος Ήβαν. Θες να πεις κάτι παρακαλώ. Intervin doar ca să mulțumesc celor care au depus eh, amendamente și Să spun că am avut o colaborare foarte bună cu Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να πω ότι ευχαριστώ τους συναδέλφους που έχουν καταθέσει τις τροπολογίες τους. Ευχαριστώ πολύ για την πολύ καλή συνεργασία με όλες τις ομάδες. Ήταν μια καλή δουλειά, μια καλή έκθεση. Οι προτάσεις ήταν επικοδομητικές πάντα. Ιδιαίτερα προβλήματα δεν είδαμε από την πλευρά τη δική μου, της κατάρτισης εκθέσεως και της επεξεργασίας των τροπολογιών. Έγιναν δεκτές όλες. Πρόκειται για μια έκθεση η οποία προχώρησε απρόσκοπτα. Και γι' αυτό θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους τους συναδέλφους για την πολύ καλή συνεργασία. Ευχαριστώ πολύ, λέει Πρόεδρος. Και ελπίζω να μπορούμε τώρα να προχωρήσουμε στη ψηφοφορία. Μην ξεχάσετε τις κάρτες για την ηλεκτρονική ψηφοφορία, γιατί είναι λίγο περίπλοκα τα πράγματα. Δεν τόσο απλά όπως μας τα εξηγεί ο Καταλήν. Κάποια σημεία θα χρειαστεί να τα κοιτάξουμε πιο μεγάλη προσοχή, γιατί είναι πιο επίμαχα από ό,τι ακούω. Γι' αυτό θέλω να είμαστε έτοιμοι και για την ηλεκτρονική ψηφοφορία. Έχετε τις κάρτες όλοι. Πολύ καλώς και ξεκινώ με την τροπολογία 22 υπέρ. Κατά. Όχι. Παρακαλώ. Ε, δεν μπορείτε να είστε και υπέρ και κατά. Υπέρ λοιπόν. Ευχαριστώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται 23 υπέρ. Κατά αποχές. Επαληθεύουμε για πρώτη φορά, αρχίζει η ψηφοφορία παρακαλώ. Το δικό μηχάνημα δεν δουλεύει. Yeah. What is closed. Πέρας 11 ψήφοι. κατά, 24 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 25 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική πρώτη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 36 υπέρ κατά αποχές. Επαληθεύουμε, αρχής ψηφοφορία παρακαλώ. 35. 36 διορθώνει η πρόεδρος. Πέρας. 14 υπέρ 6 κατά εγκρίνεται. 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 40 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 41 43 πάμε στο 43 εφόσον εγκρίθηκε υπέρ κατά αποχές Επαληθεύουμε την 43. Παρακαλώ αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρασε. Απερίφθη. 44 υπέρ. Κατά. Αποχές. Άλλη μια φορά επαληθεύουμε. 44 παρακαλώ αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. 14 υπέρ λέει η πρόεδρος, 8 κατά. 45 υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαληθεύουμε. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. 14 υπέρ 8 κατά εγκρίνεται, 46 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 54 υπέρ κατά αποχές απερίφθη, 55 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 56 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται 61 υπέρ κατά αποχές. Επαληθεύουμε. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. 9 υπέρ 13 κατά περίφθη. Σε τμήματα 62 πρώτο υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται δεύτερο υπέρ, κατά αποχές. Επαληθεύουμε το 62 δεύτερο τμήμα αρχής ψηφοφορία. Closed. Πέρας. Yeah. angenommen 11 zu 9, 12 zu 9 mit dem Kollegen χανου Χάνου Was sind wir jetzt? 62. 62 υπολογίζω και τον κύριο Τάκουλα, ο οποίο. 63, yeah. 63 τώρα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 64 υπέρ κατά αποχές επαληθεύουμε την 64 Πέρασε. χάνω δεν σε μετράω 12 υπέρ 10 κατά εγκρίνεται. 65 υπέρ κατά άποχες Α, εγκρίνεται. συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και πάω στην 72 δύο τμήματα το πρώτο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται το δεύτερο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 73 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 74 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 78 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 79 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 81-82 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 80 υπέρ όχι την 80 Ωραία, πάμε στο 83 τότε. 83 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 84 υπέρ, κατά αποχές επαληθεύουμε την 84, αρχίζει η ψηφοφορία. 10 υπέρ, 12 κατά, απερίφθη. Χάνω, δεν σε υπολογίζω. Ακόμα χειρότερα. Ε, 10, με 13 θα ήταν διαφορετικά. Ωραία, 84 ε, υπέρ, κατά 85. Εγκρίνεται. 86 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 87 υπέρ, κατά αποχές απερίφθη 88 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 89 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 90 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 92 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 93 υπέρ κατά αποχές επαληθεύουμε Πέρας της 10 υπέρ, 12 κατά απερίφθη, 94 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 95 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 96 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 98 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 99 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Η 100 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 101 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 102 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 103 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 105 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 104 υπέρ όχι. Έχει εγκριθεί. Πάμε στην 107 λοιπόν. Υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται 108 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται 109 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται 110 υπέρ κατά αποχές. Υπέρ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 124 υπέρ κατά ας επαληθεύσουμε παρακαλώ αρχής ψηφοφορία πέρας 11 υπέρ 12 κατά απερίφθη 125 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 126 ταυτόσημη 127 λοιπόν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 128 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 129 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 130 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 131 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 132 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 133 υπέρ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 Επτά υπέρ. Λοιπόν, ας επαληθεύσουμε την ε, έξι. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. 20 ψήφοι κατά. Με τρεις ψήφους υπέρ. Όπως σας είπα, απερίφθη.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 vote is closed. Πέρας. Πανηγυρικά. 24 ψήφοι υπέρ. Καμία ψήφος κατά. Καταλήν. Και στο τέλος αυτής της θητείας σου συγχαρητήρια. Σας ευχαριστούμε θερμά και περνούμε στο επόμενο θέμα. Τη αναζήτηση τη Επιτρόπου. Κάπου, κάπου σε κάποια κονία θα τη βρούμε. Μην φύγετε σε ένδειξη σεβασμού προς την Επίτροπο, παρακαλώ να είμαστε όλοι παρόντες. Μην, μην αποχωρήσετε. Α, stay here. Κοκομπού. Ach, das gehen die alle fort hier. Piotr, Boris, unglaublich.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 Es ist das letzte Treffen mit der Kommissarin für Kultur. τελευταία εμφάνιση της ε, Επιτρόπου ενώπιον μας, Επιτρόπου Αρμονδίας για τον Πολιτισμό και την Εκπαίδευση. Χαιρόμαστε πολύ, Αντρούλα, που είσαι εδώ και που μπορούμε να κάνουμε μια επισκόπηση της τελευταίας πενταετίας. Δεν ξέρω αν σας το είπα, θα το επαναλάβω πάντως. Την τελευταία πενταετία και ίσως και λίγο πιο πριν η Επιτροπή έδωσε πάρα πολλά κίνητρα σχετικά με αυτά τα οποία είναι στις ε, αρμοδιότητες μας από τη συνθήκη, έδωσε ακόμα περισσότερα κίνητρα για να προχωρήσουμε στον χώρο του πολιτισμού. Θα ήθελα λοιπόν να σε ευχαριστήσω Ανδρούλα και βέβαια όλους στο επιτελείο για την πολύ καλή συνεργασία, για την πολύ καλή όθηση με τις ανακοινώσεις, με τις συστάσεις που και εμείς μπορέσαμε να συμβάλλουμε και που ελπίζουμε ότι θα βρούνε τη θέση τους στη δουλειά των κυβερνώντων. Κυρία Επίτροπε, έχετε το λόγο. Thank you. Thank you, dear. Ευχαριστώ πολύ αγαπητή Ντόρις. Καλημέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι. Είναι μεγάλη χαρά για μένα που ε, απευθύνω το λόγο στην Επιτροπή σας, παρόλο που είναι η τελευταία φορά. Και θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω κάθε έναν και κάθε μία από εσά για τη συνεργασία σας τα τελευταία τέσσερα χρόνια, Ντόρις, όχι πέντε, εάν δεν απαντώμε. Για μας, ναι, για μας στην Επιτροπή είναι 4-4,5, για εσάς είναι πέντε χρόνια στο Κοινοβούλιο. Έστω. Τέλος πάντων, χάρη στη στήριξή σας, μπορέσαμε. Καταφέραμε, όπως είπες και εσύ Ντόρις, να πετύχουμε πολλούς από τους στόχους μας στον τομέα της εκπαίδευσης, του πολιτισμού, της νεολαίας και της άθλησης. Θα ήθελα να τονίσω κάποια από τα μεγαλύτερα επιτεύγματά μας τα τελευταία αυτά χρόνια. Πράγματι δεν καταφέραμε όλα όσα θέλαμε. Μπορούμε όμως να είμαστε περήφανοι γιατί χαράξαμε πολιτικές και δημιουργήσαμε εργαλεία τα οποία ε, θα κληρονομήσουν οι διάδοχοί μας. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια λοιπόν έκανα το παν έτσι ώστε η εκπαίδευση και ο πολιτισμός να είναι στο επίκεντρο της απάντησης που δίνει η Ευρώπη σε αυτή την πολύ μεγάλη κρίση. Περισσότερο από ποτέ οι άνθρωποι μας, οι δεξιότητες, οι ικανότητες τους είναι αυτά που θα μας επιτρέπουν να έχουμε ανάκαμψη ανάπτυξη βιώσιμη που θα περιλαμβάνει όλους, την έξυπνη ανάπτυξη που θέλουμε όλοι να δούμε. Η επένδυση στην εκπαίδευση χρειάζεται να συνεχιστεί ε, όσο περισσότερο εξηγένονται τα δημόσια οικονομικά των χωρών. Και μας ενθαρρύνει το γεγονός ότι έχουμε σημειώσει πρόοδο στους εκπαιδευτικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2020. Μέχρι το 2012 πρόπερση, το 36% των νέων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκή Ένωση φοιτούσαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και αποκτούν τις δεξιότητες και τις γνώσεις που αυξάνουν τις πιθανότητες τους να βρουν θέση απασχόλησης ικανοποιητική. Και αυτό το ποσοστό ήταν 31% στην αρχή της θητείας μας. Δηλαδή, ε, αυτή τη στιγμή προσπαθούμε και καταφέρνουμε σιγά σιγά να πετύχουμε τον στόχο μας του 40% έτσι ώστε να κλείσει το χάσμα που έχουμε με τους διεθνείς εταίρους μας. Και επιτυχάνουμε σιγά σιγά και το στόχο της ε, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, διότι ο αριθμός των μαθητών που εγκαταλείπουν το σχολείο όλο και μειώνεται. Το 2012 τα αριθμητικά στοιχεία δείχνουν μείωση ε, μέχρι το 12,7% και θα επιτύχουμε το στόχο του 10% μέχρι το 2020 ή ακόμα και νωρίτερα. Είναι σημαντική η πρόοδος αυτή, αλλά θα πρέπει να διατηρήσουμε αυτή την ορμή, τη δυναμική μας και νομίζω ότι θα το καταφέρουμε, γιατί σήμερα περισσότερο από ποτέ η εκπαίδευση είναι στο επίκεντρο της χάραξης πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτή είναι και η πιο σημαντική ε, αλλαγή που θα κρατήσει και περισσότερο σε σχέση σχέση με όλες αυτές που έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια. Είναι μια αλλαγή πιο σημαντική από τα γεγονότα και από τα νούμερα. Έχουμε θεσπίσει νέες πολιτικές, νέα προγράμματα και έχει αναγνωριστεί τελικά ότι η Ευρώπη μπορεί να κάνει τη διαφορά. Κάθε χρόνο, ε, κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, τη στιγμή κατά την οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, παρουσιάζει τις συστάσεις για στα κράτη-μέλη, πάντοτε ενισχύουμε τη στρατηγική σημασία και την τονίζουμε που έχει η εκπαίδευση ε, και η ανάγκη επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων στον τομέα της εκπαίδευσης και της παιδείας γενικότερα. Καθοδηγούμε και στηρίζουμε τις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες των κρατών μελών και έχουμε πολύ συγκεκριμένε πολιτικές όπως είναι ε, ο επανασχεδιασμός της εκπαίδευσης, το άνοιγμα της εκπαίδευσης, η διεθνοποίηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Όλα αυτά είναι δικές μας πολιτικές. Αλλά και στον τομέα του πολιτισμού έχουμε αλλάξει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουμε ε, τη βιομηχανία του θεάματος, της δημιουργίας και του πολιτισμού. Έχουμε πετύχει ένα σημείο ισορροπίας, δύσκολο να επιτευχθεί, μεταξύ της αξίας αυτής καθεαυτής που έχει ο πολιτισμός και η κουλτούρα από την άλλη, από τη μία, το ότι δηλαδή συμβάλλει στην ταυτότητά μας και από την άλλη τη σημασία που έχει από την οικονομική σκοπιά. Είναι βιομηχανίες που μπορούν να είναι επικεφαλής της καινοτομίας και να δημιουργήσουν νέες θέσεις απασχόλησης. Ε, πιστεύω όμως και θα ήθελα να είμαι ξεκάθαρη σε αυτό ότι πρέπει να παρεμβαίνει ο δημόσιος τομέας στον τομέα αυτό παρόλο που οι τέχνες και τα μίντια και ό,τι έχει να κάνει με τη δημιουργία είναι όλο πιο και πιο παγκοσμιοποιημένα και όλο και πιο ψηφιοποιημένα. Πιστεύουμε πράγματι ότι μόνη της η αγορά θα μπορούσε να είχε καταφέρει αυτό το θαυμάσιο μοσαϊκό ταινιών και τηλεοπτικών ε, προγραμμάτων το οποίο είναι τόσο ποικίλο ανε την ευρωπαϊκή επικράτεια. Φυσικά και δεν το πιστεύουμε. Η πολυμορφία λοιπόν, η ποικιλότητα, η ποιότητα, η ανεξαρτησία ε, τηλεοπτικού ε, κινηματογραφικού περιεχομένου το οποίο θα δει, χρηματοδοτείται από το δημόσιο τομέα είναι μια ευρωπαϊκή αξία και όλοι την ενστερνιζόμαστε και με περηφάνεια την υπερασπίστηκα. Ας δούμε όμως τι έχουμε κάνει τα τελευταία ε, χρόνια, τον τελευταίο χρόνο πιο συγκεκριμένα, αρχής γενομένης από τον τομέα της εκπαίδευσης. Βλέπουμε τα επίπεδα ανεργίας από τη μία σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες, τα απαράδεκτα επίπεδα ανεργία και ε, πλήττονται περισσότερο οι νέοι. Και από την άλλη πλευρά έχουμε 2 εκατομμύρια κενέ θέσει απασχόληση στην Ευρώπη και έχουμε και πάρα πολλού εργοδότε που δεν μπορούν να βρουν εργαζόμενου που να παρουσιάζουν το σωστό μείγμα δεξιοτήτων στην αγορά εργασία. Είναι λοιπόν ένα εσφαλμένο τέριασμα, αν θέλετε, μεταξύ εργοδοτών και μελλοντικών εργαζομένων. Και μέχρι το 2020, ε, σύμφωνα με τι προβλέψει μα, το 1 τρίτο των θέσεων απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα απαιτεί προσόντα υψηλή υψηλού επίπεδου, ενώ σήμερα το 1 τέταρτο ε, της, του εργασιακού δυναμικού μόνο διαθέτει τέτοιου είδους υψηλά προσόντα. Όταν παρουσίασα λοιπόν τη στρατηγική για τον επανασχεδιασμό της εκπαίδευσης πριν από ένα χρόνο, είχα ως στόχο να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη για να ανταποκριθούν σε αυτές τις προκλήσεις. Υπογράμμισα λοιπόν πόσο επίγον είναι να ε, ολοκληρώσουμε όλες αυτές τις μεταρρυθμίσεις σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης, να έχουμε το σωστό μείγμα βασικών και εγκάρσιων, αν θέλετε, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, έτσι ώστε να ενισχυθεί η απασχολησιμότητα. Να αναπτύξουμε νέες μεθόδους διδασκαλίας αλλά και μάθησης, να έχουμε νέες προσεγγίσεις ως προς τη χρηματοδότηση και τις συνεργασίες και τις εταιρικές σχέσεις. Και θα ήθελα σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω την εισηγήτριά σας, την κυρία Νεβεντάλοβα, για την έκθεσή της για τον επανασχεδιασμό της εκπαίδευσης. Γιατί η έκθεσή της ακολουθεί μια παρεμφερή προσέγγιση. Είναι μια έκθεση που εσείς εγκρίνατε, υιοθετήσατε τον περασμένο Οκτώβριο. Ο επανασχεδιασμός της εκπαίδευσης πιστεύει σημαίνει επίσης ότι πρέπει να βελτιώσουμε τη χρήση των νέων ε, τεχνολογιών στη σχολική αίθουσα. Είναι ψηφιακή εποχή την οποία διανύουμε και πολύ πρόσφατα αρχίσαμε να το ε, υιοθετούμε αυτό και στην προσέγγιση των, της διδασκαλίας και των εκπαιδευτικών μεθόδων. Μαζί με την Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Νέλη Κρούς τον περασμένο Σεπτέμβριο παρουσιάσαμε αυτή την πρωτοβουλία για το άνοιγμα της εκπαίδευσης και θέλω να συγχαρώ τον εισηγητή σας, τον κύριο Ιβάν, για την έκθεσή του. Η Επιτροπή σας την υιοθέτησε σήμερα το πρωί με ε, πολύ μεγάλη πλειοψηφία. Τον περασμένο μήνα ε, οι Υπουργοί Παιδείας της Ευρώπης υιοθέτησαν τα συμπεράσματα του Συμβουλίου. Ε, και στα συμπεράσματα αυτά αναφέρεται πράγματι και η δική μας άποψη ότι τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης δεν είναι απολύτως λειτουργικά και παραγωγικά, δεν έχουν φτάσει στο μέγιστο των ε, δυνατοτήτων τους. Πρέπει να ε, τα καταφέρουμε καλύτερα, να έχουμε το σωστό μείγμα δεξιοτήτων και προσόντων. Δεν αρκεί απλά να επεκταθεί ο αριθμός αυτών που θα φοιτήσουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Πρέπει να βελτιώσουμε την ποιότητα αλλά και αυτά τα οποία διδάσκουμε να έχουν νόημα και να είναι σχετικά. Το θέμα λοιπόν είναι να έχουν τα σωστά προσόντα, όχι μόνο περισσότερα προσόντα. Ε, πρέπει λοιπόν να έχουμε ε, καλύτερη σχέση, να ενθαρρύνουμε τη συσχέτιση και την σύσφυξη των σχέσεων μεταξύ ε, των χώρων εκπαίδευσης, διδασκαλίας και μάθησης από τη μία και των χώρων εργασίας από την άλλη. Έχουμε την Ευρωπαϊκή Συμμαχία για τη Μαθητεία. Είναι μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε το περασμένο καλοκαίρι με τον Επίτροπο Άντορ. Θέλουμε με αυτό να φέρουμε κοντά τον κόσμο της απασχόλησης και της εργασίας με τον κόσμο της εκπαίδευσης και διδασκαλίας. Έχουμε ε, ε, τις διαδικασίες της Μπολόνιας και της Κοπενχάγης. Έχουμε νέα εργαλεία ε, για να ε, αξιοποιήσουμε την πρόοδο. Αυτή τη στιγμή ε, η εστιάζουμε την προσοχή στην έρευνα ως προς την κατάταξη και δεν εξετάζουμε ιδιαίτερο στο τι γίνεται σε κάθε ένα ε, ίδρυμα στην Ευρώπη. Καμία, κανένα σύστημα κατάταξης δεν είναι τέλειο και πάντοτε υπάρχει ε, θέμα υποκειμενικότητας. Είναι χρήσιμα αυτά τα εργαλεία όμως και θα πρέπει ε, να... Ε, ε, τα χρησιμοποιούμε αναλόγως. Έχει ολοκληρωθεί λοιπόν αυτή η ευαίσθητη φάση της συλλογή δεδομένων, στην οποία έχουν συμμετέχει περισσότερα από 500 ιδρύματα σε όλο τον κόσμο και έχει ξεκινήσει η ανάλυση των αποτελεσμάτων. Τον Ιούνιο η Ελληνική Προεδρία θα οργανώσει μία διάσκεψη, ένα συνέδριο, όπου θα συζητηθούν τα πρώτα αποτελέσματα και θα ξεκινήσει ο δεύτερος γύρος ε, κατάκτης, κατάταξης. Έχουμε και το νέο πρόγραμμα, το Erasmus Sin, το οποίο μας βοηθά να εφαρμόσουμε όλες αυτές τις ε, ε, πολιτικές. Τόρη, ε, είμαι πολύ ευγνώμων σε σένα και στην Επιτροπή σας, γιατί μας βοηθήσατε να πετύχουμε αυτό το θετικό αποτέλεσμα. Χάρη στις συλλογικέ μας προσπάθειες, 4 εκατομμύρια νέοι θα έχουν την ευκαιρία να, να σπουδάσουν, να εργαστούν, να καταρτιστούν και να κάνουν εθελοντική εργασία στο εξωτερικό. Από σήμερα μέχρι το 2020 μιλούμε για 4 εκατομμύρια ανθρώπους. Το πρόγραμμα ανανεώνεται, αναβαθμίζεται και πλέον αγγίζει νέε ε, σφαίρες πολύ σημαντικέ. Με το Erasmus Συν, το Erasmus Plus, ε, θέλουμε να δείξουμε την δέσμευσή μας να προσφέρουμε ευκαιρίες αλλά και ικανότητες στους νέους ε, σε έναν κόσμο ο οποίος είναι όλο και περισσότερο κινητός θα έλεγα και πολυπολιτισμικός. Μας βοηθάει να εμπλουτίσουμε τη γλωσσική ε, πολυμορφία να ε, χρηματοδοτήσουμε τις καινοτόμες έρευνες και τις καινοτόμες μεθόδους ε, στην ε, διδασκαλία των γλωσσών, να προωθήσουμε τις περιφερειακές και μειονοτικές γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χαίρομαι ιδιαίτερος για την έκθεση του κυρίου Αλφόνσε, Αλφόνση Πέρση για την προστασία των γλωσσών εν κινδύνο. Είναι ένα νέο πρόγραμμα λοιπόν αυτό που έχουμε και όλα αυτά θα μας βοηθήσουν να αποκαταστήσουμε αυτό τις δεξιότητες με αυτά τα οποία ζητάει η αγορά. Να αποκαταστήσουμε δηλαδή το κενό που υπάρχει, να το, καλύψουμε, να το καλύψουμε και να μην υπάρχει ε, λανθασμένο, λανθασμένο τέριασμα αν θέλετε. Έχουμε 150 συμμαχίες γνώσεων που θα βοηθήσουν 1500 πανεπιστήμια και επιχειρήσεις για να είναι καινοτόμες στη διδασκαλία. Έχουμε 150 συμμαχίες για τις δεξιότητες ανατομέα και έτσι θα συνεργαστούν 2.000 εκπαιδευτικά Ινστιτούτα Κατάρτισης μαζί με επιχειρήσεις. Και σύν της άλλης το Erasmus ΣΥΝ θα δώσει νέα ενέργεια, νέα πνοή ε, στους νέους σε καιρούς υψηλών ποσοστών ανεργίας και θα βοηθήσει τους νέους που έχουν αποχωρήσει από το σύστημα. Κάτι το οποίο μας ανησυχεί ιδιαιτέρως. Στην αρχή ορισμένοι είχαν επιφυλάξεις για το πρόγραμμα αυτό το νέο. Όμως το τελικό αποτέλεσμα είναι καλό γιατί με το Erasmus Sinner θα, θα αποκτήσει περισσότερη ορατότητα το πόσο μπορεί να βοηθήσει η άτυπη, η μη επίσημη μάθηση και διδαχή. Έτσι μπορεί κανείς να αποκτήσει πολύ σημαντικές δεξιότητες ακόμα και αν βρίσκεται εκτός σχολικής αίθουσες. Ε, θα έχουμε αυξημένη χρηματοδότηση για τον εθελοντισμό, για την εργασία της νεολαίας η οποία θα αποκτήσει εμπειρία. Θα μάθουν και θα ε, γνωρίσουν οι νέοι άνθρωποι περισσότερα για την αξία ε, της αγωγής του πολίτη, της συμμετοχής τους στην ε, ζωή, στην κοινωνία. Για όλους αυτούς τους λόγους θα ήθελα λοιπόν να υπενθυμίσω τη σημασία της έκθεσης του κυρίου Παπα-Νικολάου, να τον συγχαρώ και να τον ευχαριστήσω για την υιοθέτηση της έκθεσης αυτής πέρσι για την νεολαία, για τους νέους. Ως προς την άθληση, νομίζω ότι προσπαθήσαμε να αφιερώσουμε αρκετό χώρο στην άθληση στο νέο αυτό είναι πολύ σημαντικό όλο αυτό. Για πρώτη φορά τα αθλήματα θα έχουν ε, ε, το δικό τους εργαλείο χρηματοδότησης ε, στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εδώ έρχεται και η έκθεση φύσας για την ευρωπαϊκή διάσταση στον αθλητισμό. Which I know is... Ας έλθω τώρα στα θέματα του πολιτισμού, τα οποία σας ενδιαφέρουν φυσικά ή ιδιαίτερα όπως ενδιαφέρουν και εμένα. Εδώ κάναμε αρκετές, ε, προωθήσαμε αρκετές νέες ιδέες στον τομέα της ε, δημιουργικότητας και προστατεύοντας ε, την ποικιλότητα, την πολιτιστική. Αυτό δίδει κίνητρα για καινοτομίες, δίδει κίνητρα για την επιχειρηματικότητα. Στη στρατηγική που παρουσίασα για την προώθηση του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα, επέμεινα ότι ο πολιτισμός έχει τεράστιο δυναμικό όχι μόνο για την ανάπτυξη και νέες θέσεις απασχόλησης αλλά για να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών στο ευρωπαϊκό όραμα και να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη ανάμεσα στην οικονομία και την κοινωνία. Είμαι ευγνώμων για την υποστήριξή σας στη στρατηγική αυτή και ευχαριστώ κυρίως την κυρία Σάντσες Σμιτ για την εξαιρετική της έκθεση σε αυτόν τον κλάδο. Φυσικά οι επιτυχίες μας εκμεταλλεύτηκαν την πολιτιστική μας ικανότητα και εξαρτάται φυσικά από τη διασφάλιση της επαρκούς χρηματοδότησης της δημιουργικότητας και ενός διακανονιστικού περιβάλλοντος όπου μπορεί να βοηθήσει να ανθίσει ο πολιτισμός. Οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες πολιτισμού έδειξαν επανειλημμένα ότι ενσωματώνοντας τον πολιτισμό και τις τέχνες στις μακρόπνοες αναπτυξιακές του στρατηγικές μπορούν να δημιουργήσουν νέες θέσεις απασχόλησης. Αυτό είναι κάτι που θα μας βοηθήσει ε, για το δυναμικό μέλλον μας. Να ευχαριστήσω εδώ τον κύριο Σκουρία για την έκθεσή του για την ανανέωση των Ευρωπαϊκών Πρωτευουσών Πολιτισμού. Η υποστήριξή σας κατά τη διάρκεια των δύσκολων διαπραγματεύσεων ήσαν πολύτιμες και γνωρίζω ότι η Επιτροπή σας ε, στήριξε μια συμβιβαστική λύση του Φεβρουάριο, τον Φεβρουάριο που θα μας επιτρέψει να ολοκληρώσουμε με επιτυχία. Επίσης ε, και ε, το Ευρωπαϊκό Σήμα για τον Πολιτισμό. Ευχαριστώ και την κυρία Παλιαδέλη εδώ και πράγματι βλέπουμε ήδη τους πρώτους καρπούς των προσπαθειών μας. Ε, την Άνοιξη θα προτείνω και μια νέα πρωτοβουλία η οποία θα ανοιχνεύσει το πόσο ο πολιτισμός συνεισφέρει στις οικονομίες και τις κοινωνίες μας και πόσο στηρίζει το ευρωπαϊκό πρόγραμμα και όραμα. Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατανοώντας τον ε, πολιτισμό, την πολιτιστική κληρονομιά και να ξεκινήσουμε και μία συζήτηση με τις κοινωνίες για το πώς θα συνεργαστούμε καλύτερα. Και έχουμε επίσης ξεκινήσει και το νέο πρόγραμμα για την Δημιουργική Ευρώπη με ένα προϋπολογισμό 1,5 δις, 9% περισσότερο από πέρυσι. 9% σε μια φάση όπου ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός έχει μειωθεί Πολύ συχνά όπως γνωρίζετε το ξεχνά ο κόσμος αυτός και λέει ότι είναι μικρά η αύξηση, αλλά είναι τεράστια όταν όλα τα άλλα μειώνονται. Χάρη στη στήριξή σας μπορούμε να στηρίξουμε ακόμα περισσότερο ε, τους καλλιτέχνες, τον κινηματογράφο και τις μεταφράσεις της λογοτεχνικές, ενισχύοντας την διεθνή τους ανταγωνιστικότητα και διατηρώντας την ποικιλότητά μας. Στηρίζουμε συνεχώς λοιπόν τον πολιτισμό και την δημιουργία. Ε, εγώ ζήτησα από τα κράτη-μέλη και έστειλα επιστολές προσωπικά σε όλους τους υπουργούς, τους υπεύθυνους για τα τα ταμεία και την ανάπτυξη να στηρίξουν τον πολιτισμό σαν τμήμα μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής περιφερειακής ανάπτυξης. Επέμεινα ότι τα διαφθορτικά ταμεία βρίσκονται εκεί για να στηρίξουν και τις ευφυείς επενδύσεις. Την άνοιξη πάλι λοιπόν, ε, μάλλον ε, καλύτερα νομίζω ότι σήμερα καταλαβαίνουμε ότι το θέμα της χρηματοδότησης του πολιτισμού είναι πολύ σημαντικό θέμα αυτοί που ασχολούνται με τον πολιτισμό έχουν ανάγκη από ειδικέ μορφές χρηματοδότησης από, δημόσιες, από δημόσιους πόρους και ιδιωτικούς πόρους. Γι' αυτό ακριβώς και με το πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη, Creative Europe, θα αντιμετωπίσουμε κατά μέτωπον αυτές τις προκλήσεις. Ιδιαίτερα σε αυτή την εποχή της αυστηρής λιτότητας οι προσπάθειές μας φαίνονται ξεκάθαρα και ευχαριστώ και την κυρία Κώστα η οποία σαν εισηγήτρια βοήθησε για να ολοκληρωθεί η διαδικασία με επιτυχία. Αν δούμε λοιπόν λίγο προς τα πίσω και εξετάσουμε όλα αυτά τα προγράμματα, το Erasmus Sin, το Creative Europe και τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, βλέπουμε ότι υπάρχει πραγματικά μια προσδοκία το όραμά μας να γίνει πραγματικότητα, το όραμα μιας Ευρώπης ανοιχτής, δεκτικής, με εμπιστοσύνη που θα βοηθήσει τους νέους. Μια Ευρώπη η οποία είναι ανοιχτή και στους πολίτες της αλλά και στους γείτονες και στον υπόλοιπο κόσμο. Χάρη και στην δική σας προσπάθεια, σκληρή προσπάθεια, πετύχαμε αυτά τα ικανοποιητικά αποτελέσματα. Σας ευχαριστώ για μια ακόμη φορά για αυτήν την τελική δυνατότητα να μοιραστώ κάποιες σκέψεις μαζί σας. Θέλω να ευχαριστήσω και τις αντιπροέδρους, ιδιαίτερα την κυρία Τρούπελ και τον κύριο Λόκεγκάρντ με τους οποίους συνεργάστηκα στενότατα. Φυσικά οι τελευταίες λέξεις μου αφορούν την προεδρό σας. Θα ήθελα εδώ να αποτίσω φόρο τιμής σε σένα, Ντόρις. Δεν είχα τη δυνατότητα να το κάνω χθες, νομίζω ότι τώρα είναι καταλληλότερη στιγμή. Ε, η πραγματικά διακριτή σταδιοδρομία σου σε αυτό το κοινοβούλιο και σε αυτή την επιτροπή σφράγισε την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις πολιτικές της. Μπορείς να είσαι υπερήφανη για την κληρονομιά σου και σου εύχομαι κάθε προσωπική επιτυχία στο μέλλον. Thank you very much, dear. Ε, Ευχαριστούμε πολύ, αγαπητή Ανδρούλα. Και τώρα παρακαλώ τους συναδέλφους να λάβουν το λόγο. Κυρία Κάμερεβερτ, ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ πολύ κυρία Επίτροπε που είχατε την καλοσύνη να μας παρουσιάσετε τόσο ευρία επισκόπηση των όσων έχουμε από κοινού επιτύχει τα τελευταία 4,5-5 χρόνια. Θα ήθελα πάντως να είμαι... να ε, κατεβάσω λίγο τους τόνους το ΣΥΠΗΝ για να πω ότι το πρόγραμμα Erasmus Plus είναι και να πω ότι πέρασε αρκετό καιρό εδώ στην Επιτροπή και χρειάστηκε να περιμένουμε μέχρι ότου μπορέσουμε να πείσουμε την Επιτροπή ε, για να δεχθεί τις δικές μας προτάσεις ότι είναι οι καλύτερες και οι πιο σωστές. Καταφέραμε βεβαίως να θέσουμε σε κίνηση καλά προγράμματα, αναμφίβολα. Στις 12 Δεκεμβρίου και με μεγάλη χαρά μπορέσαμε να εγκρίνουμε το, το πρόγραμμα Guide για το Erasmus Plus. Σήμερα 18 Μαρτίου και αυτό προκύπτει από ένα τηλεφώνημα με την Επιτροπή εχθές. Σήμερα 18 Μαρτίου έχουμε και άλλες γλωσσικές εκδόσεις για τις ε, προγραμ... Ε, δεν έχουμε ακόμη άλλες γλωσσικές εκδόσεις πριν της αγγλικές για το Erasmus Plus. Και μαθαίνουμε λοιπόν ότι Τώρα μπορεί να εμφανιστεί μια γαλλική και γερμανική εκδοχή του κειμένου, η οποία τώρα θα πάει στις ε, οικίες εθνικές αντιπροσωπείες Παρίσι-Γερμανία για επαλήθευση της γλώσσας Φαντάζομαι όμως ότι δεν είναι καν αρμόδιες οι εθνικές αντιπροσωπείες για κάτι τέτοιο. Έτσι, κείμενο της Επιτροπής είναι. Η Επιτροπή πρέπει να έχει την ευθύνη για τη μετάφραση και την επαλήθευση της μετάφρασης. Και ότι ίσως σε 14 μέρες ενδέχεται αυτές οι δύο γλωσσικές εκδόσεις να είναι επίσημες. Αλλά και αυτό πάλι με πολύ εντατικούς ρυθμούς μας λένε. Για δε τις λοιπές ε, γλωσσικές εκδόσεις δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί πότε θα είναι διαθέσιμες. Γιατί να χρειάζεται τόσο πολύ. Έστω είναι ογκώδες το έγγραφο, έστω δεν έχετε κόσμο όμως. Μα η Επίτροπος η αρμόδια για την πολυγλωσία μπορεί και όταν ξέρει και ότι η, Επιτροπή δική μας πάντοτε δίνει πολύ μεγάλη σημασία και ότι σε τελευταία ανάλυση και άλλες γενικές ε, διευθύνσεις βλέπουμε να έχουν ανοίξει διαβουλεύσεις μόνο στα αγγλικά έστω. Άλλες ναι, αλλά στο δικό σας τον τομέα που ασχολείται με την πολυγνωσία, να βλέπουμε τέτοιες καθυστερήσεις προς τις διαφορετικές γλωσσικές εκδόσεις και το Creative Europe επίσης. Οι κατευθυντηρίες γραμμές για το τομέα της, ε, του πολιτισμού θα έπρεπε Έστω μπορεί να υπάρχουν στα γαλλικά, αγγλικά, γερμανικά γλώσσε εργασία, αλλά πάλι θα έπρεπε να ξέρουμε πότε θα είναι διαθέσιμε οι λοιπέ εκδόσει. Και το media επίση. Μόνο στα αγγλικά δυστυχώ. Λοιπόν, στον τομέα αυτό, με όλη τη στράτευση, με όλες τις προσπάθειες, τις ε, ταινιούλες που βγάζουμε στην ιστοσελίδα της Επιτροπής και που θεωρώ ότι θα έχουν σχετικά περιορισμένη προσθέμενη αξία σε σχέση με το θέμα που εγώ θίγω. Νομίζω ότι λάθος είναι οι προτεραιότητες που, που δίνεται. Και γι' αυτό παρακαλώ κατεπηγόντως να και στο πλαίσιο των χρονικών περιθωρίων που έχετε για τις θητείες σας, να πιέσετε όσο το ταχύτερο δυνατό οι προγραμματικές κατευθυντήριες γραμμές να είναι διαθέσιμες σε όλες τις γλώσσες, γιατί αυτό νομίζω ότι αποτελεί και όρο τον νόμο κάνει για την επιτυχία των προγραμμάτων. Για να μπορούν οι πολίτες στις χώρες μέλη να ενημερώνονται στη γλώσσα τους για το ποιες δυνατότητες προσφέρει το Erasmus Plus, για το ποιες δυνατότητες προσφέρει το Creative Europe και ούτω καθεξής. Το Creative Europe μάλιστα θα ήθελα να το θέξω ακόμη για, με μια φράση. Έχουμε την εντύπωση με τις κατευθυντήρε γραμμές για το Creative ε, Europe ότι δεν ε, φαίνεται να έχει ληφθεί σοβαρά υπόψη το τι συμφώνησαν το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο, διότι η έννοια της προστέμενης ευρωπαϊκής αξίας, για την οποία εμείς αγωνιστήκαμε πολύ και έχουμε δώσει μεγάλη σημασία, για τις κατευθυντήριες γραμμές στον χώρο του πολιτισμού ιδιαίτερος, Νομίζω ότι εμφανίζεται μόνο μία φορά και μάλιστα παρεμπιπτόντω σε μια δευτερεύουσα θέση. Εν πάση περιπτώσει, θα ήθελα να εμφανίζεται πολύ πιο ξεκάθαρα. Γιατί αυτό το οποίο έχουμε από κοινού αποφασίσει πρέπει να βρίσκεται μέσα στις κατευθυντήριες γραμμές για τα προγράμματα και να εμφανίζεται ξεκάθαρα. Ευχαριστώ πολύ, Μαγιτάρες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επίτροπε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την στήριξή σας στις προσπάθειες τις οποίες από κοινού κάναμε και να ευχαριστήσω φυσικά και την Τόρις για την προεδρία της και για τη δραστηριότητα της σε όλες αυτές τις προσπάθειες. Να αναφερθώ σε δύο σημεία εδώ, εκπαίδευση και πολιτισμός. Πρώτα πολιτισμό. Χαίρομαι γιατί η προσπάθεια την οποία κάναμε μέχρι τώρα ε, βοήθησε τα κράτη-μέλη να κατανοήσουν το δυναμισμό που κρύβει ο πολιτισμός στη Γαλλία ιδιαίτερα υπήρξε μια έκθεση η οποία έδειξε ξεκάθαρα και με αριθμητικό τρόπο τον δυναμικό, το οικονομικό του τομέα του πολιτισμού. Ο πολιτισμός δεν είναι κάτι που έχει σαν αποκλειστικό στόχο μια μικρή ελίτ, αλλά είναι κάτι που δημιουργεί θέσεις απασχόλησης, βοηθά τους νέους, και σας ευχαριστώ για τα λόγια σας ότι πέραν και του οικονομικού δυναμικού ο πολιτισμός θα βοηθήσει την ανάκτηση της εμπιστοσύνης των πολιτών στην Ευρώπη. Τώρα για το διατλαντικό, για το μάλλον σύμφωνο αναφερθήκατε στα θέματα της πολιτιστικής εξέρεξης, ε, αναφερθήκατε στα θέματα των ραδιοτηλεοπτικών παραγωγών, όλα αυτά σε σχέση με τις συμφωνίες αυτές. Ποια είναι η γνώμη σας. Δεν έχουμε πάρα πολλές πληροφορίες σχετικά με τις διαπραγματεύσεις. Τι ακριβώς θα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον τομέα που μας ενδιαφέρει στις συζητήσεις αυτές. Η στρατηγική της Επιτροπής δεν ήταν απόλυτα συμβατή με τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο παρελθόν. Εμείς εμένουμε επίτροπε στην πολιτιστική εξαίρεση. Έχουμε εγγυήσει ότι οι ΙΠΑ δεν θα επανέλθουν και θα αμφισβητήσουν το θέμα αυτό το τόσο σημαντικό για μας. Τώρα, δεύτερον, είναι το ΦΠΑ online. TVA online. Ε, ξέρετε ότι εγώ επιμένω να παραμείνει χαμηλό το ποσοστό επιβολή σε ό,τι αφορά τον πολιτισμό. Η Ευρωπαϊκή νομοθεσία επιτρέπει αποκλήσεις, επιτρέπει εξαιρέσεις. Πού βρίσκονται λοιπόν οι διαπραγματεύσεις. Αναμένουμε μια ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα μειωμένα ποσοστά σύντομα μετά από την ολοκλήρωση των μελετών επιπτώσεων. Έχετε κάποιες πληροφορίες για τις εξελίξεις αυτές στον τομέα της εκπαίδευσης. Συμφωνώ απολύτως επίτροπε με την ανάλυση σας. Έχουμε ανάγκη για ένα καλό συντονισμό ανάμεσα στα εκπαιδευτικά συστήματα, την καινοτομία και την κινητικότητα τον Φεβρουάριο του 2004 το δημοψήφισμα των Ελβετών εν μέρη έθεσε σε αμφισβήτηση θα έλεγα ε, και μπορεί να προκαλέσει κάποια προβλήματα στην αρχή της ελεύθερης διακίνησης των πολιτών ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελβετία φαίνεται ότι θα πρέπει να συζητήσουμε και να διαπραγματευτούμε εκ νέου με τους Ελβετούς για τα θέματα της κινητικότητας. Ποια είναι η άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν έχω άλλες ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Ε, Σαντιάγο και Να και μετά θα δώσουμε μια ευκαιρία. Σαντιάγο πρώτα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επίτροπο, την αγαπητή κυρία Ανδρούλα Βασιλείου, για την παρουσίαση που μας έκανε. Θα ήθελα επίσης να σας συγχαρώ για τη διεραστηριότητά σας αυτά τα τέσσερα ή πέντε χρόνια. Πέντε για εμάς, τέσσερα για σας. Για το ότι πάντοτε ήσασταν κοντά μας. Κάθε φορά που χρειάστηκα να σας μιλήσω, με υποδεχθήκατε, ε, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και με πολύ μεγάλη προσοχή με ακούσατε. Θέλω να σας συγχαρώ για την αύξηση του προπολογισμού επίσης που πετύχατε σε όλους τους τομείς ε, του χαρτοφυλακίου σας, κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό ε, σε περίοδο κρίσης. Μια εποχή κατά την οποία περικόπτονται οι προϋπολογισμοί παντού. Όμως τα θέματα που απασχολούν τις Επιτροπή μας έτυχαν προϋπολογισμό ο οποίος όχι μόνο δεν μειώθηκε αλλά αυξήθηκε κιόλα. Και θα ήθελα να κάνω μια μικρή αναφορά στην άθληση, στα αθλήματα, κάτι το οποίο μας ενδιαφέρει ιδιαίτερος και κάτι το οποίο είδαμε ότι ενδιαφέρει ιδιαίτερα και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τη διάρκεια της δικής σας θητείας, κυρία Βασιλείου. Αυτό λοιπόν που θα ήθελα να πω είναι το εξής. Η έκθεση που ψηφίσαμε εδώ και θετήσαμε με μεγάλη πλειοψηφία, στην οποία αναφερθήκατε προηγουμένως, θα ήθελα να μην παραμείνει σε κάποιο σιρτάρι. Ξέρω ότι δεν είναι νομοθετικού χαρακτήρα έκθεση, ωστόσο περιλαμβάνει πάρα πολλές χρήσιμες ιδέες που θα έπρεπε να προωθηθούν περαιτέρω. Κυρίως μιλώ για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλημάτων Έχουμε μιλήσει γι' αυτό και εάν δεν απατώμε τον Ιούνιο θα γίνει μια μεγάλη συνάντηση με τους ε, διαφόρους συμμετέχοντες για τα θέματα της άφλησης και των αθλημάτων για να προωθηθεί όλο αυτό η, η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα αθλημάτων και άθλησης και θα μπορούσε να οργανωθεί η 1η του Σεπτέμβριου του 2015. Θα ήθελα περισσότερα ε, στοιχεία γι' αυτό. Ευχαριστώ. Η κυρία Τρίου και θα ακούσουμε τις πρώτες απαντήσεις. Ευχαριστώ Ντόρις, ευχαριστώ Επίτροπε Βασιλείου για την ομιλία σας, για την ε, επισκόπηση. Όσον αφορά το πρόγραμμα Creative, Creating Europe, ξέρετε ότι έχουμε συζητήσει ιδιαίτερως το θέμα του τι θα μπει στη νέα δομή, τη συνεργασία μεταξύ των ε, ε, γραφείων επικοινωνίας και των σημείων επαφής και γι' αυτό θα ήθελα να μου πείτε πόσο έχει προχωρήσει αυτή η υπόθεση γιατί με ενδιαφέρει πολύ η ορατότητα των προγραμμάτων και θα πρέπει το Media Desk να το ξεχωρίσουμε από το ε, Cultural Content Desk. Ε, πείτε μας λοιπόν πόσο έχει προχωρήσει και τι περιμένετε ότι θα γίνει στο εγγύς μέλλον στον τομέα αυτό και επίσης στην ε, τρέχουσα αυτή περίοδο είχαμε την προετοιμασία των ε, πολιτιστικών εξωτερικών σχέσεων. Θα έχουμε τον Απρίλιο μια διάσκεψη. Θα ήθελα όμως να ακούσω και από εσά τις ιδέες σας για το τι περιμένετε σε αυτόν τον τομέα της πολιτικής, για τον εξωτερικό ρόλο του πολιτισμού. Και θα ήθελα να αναπτύξετε περισσότερο αναλυτικά τις ιδέες σας στον τομέα αυτό. Αντρούρα, ένα λεπτό μόνο, επειδή πρέπει ο συνάδελφος να ή συνάνθρωπο να πάει στην Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού για να ψηφίσει. Μια πολύ στομή ερώτηση, γιατί βέβαια και οι υπόλοιποι θα πρέπει να μιλήσουν. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ψηφίζουμε την απαλλαγή τη Επιτροπής και γι' αυτό πρέπει να σπεύσω, να επιστρέψω. Έχω μια ερώτηση, λοιπόν, για μία από τις δικές μου προτάσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρόταση για το 2017 να χαρακτηριστεί έτος της επιχειρηματικότητας για να υποστηρίξουμε την επιχειρηματικότητα και το πνεύμα του επιχειρήν στους νέους και να προαγάγουμε με περισσότερα μέσα και πρακτικά παραδείγματα των αγώνα κατά της ενεργείας των νέων. Η κατάρτιση βέβαια και η εκπαίδευση έχουν πολύ σημαντικό ρόλο στην υπόθεση αυτή. Ποια είναι η θέση σας για την πρόταση αυτή το 2017 να ανακηρυχθεί Ευρωπαϊκό Έτος της Επιχειρηματικότητας ή του επιχειρήν. Ευχαριστώ. Την απάντηση θα την λάβεις αργότερα, μια και πρέπει να φύγεις για την ψηφοφορία, θα ενημερωθείς μετά. Παρακαλώ τους κλητήρες μας, με ακούτε, οι κύριοι κλητήρες. Αν, θέλετε να συνομιλείτε, σας παρακαλώ πολύ να βγείτε από την αίθουσα. Um, Ευχαριστώ πολύ. Ας ξεκινήσω από τη μετάφραση. Να μην ξεχνούμε ότι αυτή τη χρονική στιγμή όπου έχουν υιοθετηθεί και εγκριθεί όλα αυτά τα προγράμματα, η πρόκληση για την Γενική Διεύθυνση ε, με τη Μεταφραστική Υπηρεσία είναι τεράστια. Δεν συνηθίζει να πρέπει να μεταφράζει τεράστια τεύχη εγγράφων, ε, τεράστιους όγκους μεταφραστικού έργου. Δεν μιλούμε για τα δικά μας προγράμματα, ε, προγράμματα μόνο. Υπάρχει και το πρόγραμμα Citizens, υπάρχει και το Ορίζοντας για το 2020, πάρα πολλά και διαφορετικά πράγματα. Και πρέπει η Γενική Διεύθυνση αυτή να διεκπαιρεώσει αυτό το τεράστιο μεταφραστικό έργο ταυτοχρόνως, γιατί όλα εγκρίθηκαν την ίδια στιγμή. Ας σας πω όμως λίγα λόγια για το δικό μας πρόγραμμα. Η πρώτη προκήρυξη υποβολής προτάσεων για το Εράσμους Συν δημοσιεύθηκε σε όλες τις επίσημες γλώσσες. Η διαδικτυακή τοποθεσία για το Erasmus είναι μεταφρασμένη και διαθέσιμη σε όλες τις επίσημες γλώσσες. Έχουμε δώσει εντολή στις ε, σχετικές υπηρεσίες να δίνουν πληροφορίες και εξηγήσεις στους ενδιαφερομένους όσους θέλουν, όσοι θέλουν να υποβάλουν και αυτά τα στοιχεία να τα δίνουν στην αντίστοιχη γλώσσα του καθενός. Το πρόβλημα είναι με τον οδηγό ε, του προγράμματος, ένα πολύ μακροσκελές κείμενο 300 σελίδων. Μεταφράζεται. Ε, έχουμε τώρα ολοκληρώσει την αγγλική, τη γαλλική και τη γερμανική εκδοχή του κειμένου και όλες οι άλλες γλώσσες ε, θα ε, μεταφραστεί σε όλες τις άλλες γλώσσες ε, όσο πω. Και ελπίζω ότι σύντομα θα έχετε τη μετάφραση σε όλες τις γλώσσες. Δεν είναι δηλαδή επειδή εμείς υποτιμούμε τη σημασία των άλλων γλωσσών. Όχι, καθόλου. Όμως είναι θέμα εργασιακού δυναμικού. Δεν γίνεται δεν έχουμε αυξήσει ε, τους πόρους μας για την ε, γενική διεύθυνση που έχει τη μεταφραστική υπηρεσία. Αντιθέτως, μειώνουμε λόγω περικοπών το προσωπικό, ενώ αυξάνεται το μεταφραστικό έργο. Είναι τεράστιος ο όγκος της δουλειάς και πρέπει να τα φέρουμε σε πέρας. Έχουμε και εμπορικές συμφωνίες, πολλά και διάφορα πράγματα που έρχονται και κατακλείζουν τη μεταφραστική υπηρεσία. Να μην υποτιμούμε την αξία της δουλειάς, της γενικής αυτής διεύθυνσης. Ε, κάνουν ένα έργο ε, πολύ μεγάλο, πρέπει να δείξουμε κατανόηση σε πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες. Τώρα, ως προς την ευρωπαϊκή Προσθεθέμενη αξία στο πρόγραμμα για την δημιουργική Ευρώπη. Πιστεύω ότι και στο πρόγραμμα και στον οδηγό πάρα πολλά σημεία υπογραμμίζουν ποια είναι πραγματικά η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Ε, η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών αυτή είναι μια προστιθέμενη αξία αυτή καθεαυτή, γιατί με κανέναν άλλο τρόπο οι επαγγελματίε στον τομέα των τεχνών και των πολιτισμών δεν μπορούν να συνεργαστούν με άλλους συναδέλφους τους και να παράξουν ένα αποτέλεσμα τόσο σημαντικό ε, για την Ευρώπη. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν μόνο και αυτό ε, έχει μια προστιθέμενη αξία από μόνο του και νομίζω ότι το εκτιμούν όλοι ιδιαιτέρω. Τώρα, ως προς τον οικονομικό αντίκτυπο του πολιτισμού και της κουλτούρας. Είναι πολύ σημαντικό να τον έχουμε υπόψη μας αυτό, αυτόν, ειδικά σε καιρούς κρίσης. Να σας πω ότι πριν από ένα μήνα με το Κοινό Κέντρο Ερευνών ξεκινήσαμε ένα project ένα πρόγραμμα ερευνητικό για να κάνουμε συνεχώς έρευνες και να καταλήξουμε σε στοιχεία απτά συγκεκριμένα για το πόσο μεγάλη αξία έχει ο πολιτισμός στην οικονομία μας, για το πόσο μεγάλος είναι ο αντίκτυπος του πολιτισμού με όρους αξίας οικονομικής στις κοινότητές μας και στις κοινωνίες μας. Χρειάζονται τέτοια στοιχεία απτά όσοι είναι υπεύθυνοι για τη χάραξη της πολιτικής οι ηθήνοντες για να ε, φέρουν την κουλτούρα και τον πολιτισμό στο προσκήνιο. Τώρα, η πολιτιστική εξαίρεση. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι είναι κάτι που στηρίζω, που στήριζα εξ αρχής. Είχε αποκλειστεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και τώρα λοιπόν οι διευθύνσεις ε, τις οποίες εποπτεύω παρακολουθούν εκ του και τι ε, συζητήσει κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Δεν είμαστε μέρος της διαπραγματευτικής ομάδας, αλλά είμαστε παρόντες. Ανά πάσα στιγμή παρατηρούμε και διασφαλίζουμε ότι ούτε με άμεσο τρόπο, ούτε με έμεσο τρόπο ε, δεν θα τεθεί το θέμα της πολιτιστικής εξαίρεσης της διαπραγματεύσης. Τώρα, ως προς την Ελβετία, πράγματι ήταν πολύ ατυχές αυτό το συμβάν. Ξεκινήσαμε τις διαπραγματεύσεις με τις ελβετικές αρχές τον Δεκέμβριο και λέω δυστυχώς λόγω του δημοψηφίσματος, διότι λόγω του δημοψηφίσματος ε, έπρεπε να διακόψουμε τις διαπραγματεύσεις. Περιμένουμε διευκρινήσεις από πλευράς Ελβετών για να δούμε πώς θα εφαρμόσουν την απόφαση του δημοψηφίσματος και να δούμε πώς μπορούμε να συνεργαστούμε με την Ελβετία. Δεν θα πλήξει αυτό με κανένα τρόπο ε, την τρέχουσα πανεπιστημιακή ε, χρονιά, ε, εκπαιδευτικό έτος 2013-2014 γιατί όλα αυτά έχουν αποφασιστεί εκ των προτέρων με τα προηγούμενα προγράμματα. Είμαστε λοιπόν ε, σε αναμονή ε, διευκρινήσεων από τους Ελβετούς. Τώρα για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Άθλησης και Αθλημάτων. Όπως γνωρίζετε κύριε Φίσα, Ήδη έχουμε οργανώσει μια συνάντηση μεταξύ εμπλεκόμενων φορέων για να υπάρξει ανταλλαγή καλών πρακτικών, για να πάρουμε πληροφορίες και ε, να δεχθούμε προτάσεις από τους εμπλεκόμενους φορείς για το πώς θα μπορούμε να οργανώσουμε καλύτερα αυτή την εβδομάδα. Έχουμε κάνει λοιπόν όλη αυτή τη δουλειά και στις 11 Ιουνίου θα έχουμε αυτή την πολύ μεγάλη ε, διάσκεψη, αυτό το ε, συνέδριο στο οποίο θα κληθούν να αναλάβουν δεσμεύσεις οι εμπλεκόμενοι φορείς και χρειαζόμαστε τη δέσμευσή τους, την ενεργή, την ουσιαστική ε, πριν από την έναρξη της διοργάνωσης και πιστεύουμε πράγματι ότι η πρώτη εβδομάδα άθλησης θα λάβει χώρα το Σεπτέμβριο του 2015. Τώρα, ως προς το Media Desk, Έχουμε ε, τη θηρίδα, το τέσκε για τη Δημιουργική Ευρώπη σε πολλά κράτη-μέλη. Σε ορισμένα κράτη-μέλη αποφάσισαν να έχουν θηρίδα για τα μίντια και θηρίδα για τον πολιτισμό ξεχωριστή. Ένα τέσκε, ένα γραφείο υποδοχής. Το κάθε κρατος μέλος θα αποφασίσει αν θα έχει ένα ή δύο. Ως προς το επιχειρηματικό πνεύμα, την επιχειρηματική δραστηριότητα, είναι μία από τις δεξιότητες που χρειάζονται όλοι ανεξαιρέτως οι νέοι μας ε, στην Ευρώπη. Να έχουν δηλαδή την αίσθηση του επιχειρήν. Ε, γιατί αυτό είναι που μας θέτει σε μειονεκτική σχέση σε σχέση με τις ΙΠΑ ή την Ιαπωνία. Πρέπει δηλαδή να ξεκινήσουμε την εκπαίδευση στο επιχειρήν από πολύ νεαρή ηλικία. Να διδάξουμε στους νέους πώς θα αναλάβουν κινδύνους και ρίσκα. Γιατί χωρίς αυτή την οτροπία δεν θα είναι σε θέση να γίνουν επιχειρηματίες στην Ευρώπη. Και το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Καινοτομίας και Τεχνολογίας είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα ε, του τρόπου με τον οποίο ε, το επιχειρηματικό πνεύμα, η επιχειρηματική κουλτούρα αν θέλετε, ε, οδηγεί σε αποτελέσματα. Ταυτόχρονα με την εκπαίδευση στον εκάστοτε τομέα. Σε αυτή τη χρονιά λοιπόν του επιχειρήν θα έχουμε καλά αποτελέσματα ε, ελπίζω και θα ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη έτσι ώστε να συμπεριλάβουν τη διδασκαλία στις μεθόδους επιχειρήν και στην οτροπία του επιχειρήν από την πολύ νεαρή ηλικία μέχρι και την τριτοβάθμια ε, εκπαίδευση. Τώρα, οι πολιτιστικές εξωτερικές σχέσεις. Το είπατε και εσείς πράγματι, θα γίνει μια ε, πολύ μεγάλη διάσκεψη για το θέμα αυτό. Συνεργαζόμαστε ε, στενά με τις σχετικές υπηρεσίες, ε, τα σχετικά τμήματα από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Θέλουμε να καλλιεργήσουμε τη σωστή νοοτροπία σε όλα τα κράτη-μέλη. Να συμπεριλάβουν δηλαδή τη διάσταση του πολιτισμού και της κουλτούρας στις εξωτερικές σχέσεις του κάθε ενός. Και έχουμε συστάσεις στα κράτη-μέλη και έχουμε και ένα πιλωτικό πρόγραμμα με την Κίνα, αλλά δεν θα είναι η Κίνα η μόνη περίπτωση. Δουλεύουμε και ε, με τη Βραζιλία πάνω σε αυτό το θέμα και ελπίζω ότι αυτό ε, τελικά θα γίνει μόνιμο χαρακτηριστικό των εξωτερικών σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο μέλλον. Ευχαριστώ. Η κυρία Φερχαέν. Ναι, καταρχάς ευχαριστώ πολύ και για την επισκόπηση των τελευταίων ετών και των πρωτοβουλειών στον τομέα του πολιτισμού. Σε δύο σημεία έχω ακόμα να ρωτήσω. Καταρχάς για την εκπαίδευση, για την παιδεία τα τελευταία χρόνια με την κρίση αντιληφθήκαμε ότι πολλοί νέοι δεν μπορούν να βρουν μια θέση εργασίας και πρέπει να βρεθούν αντιμέτωποι με το δίλημα της ε, εξασφάλισης μιας θέσης εργασίας, της εκκίνησης δηλαδή στον επαγγελματικό βίο. Άρα το ζήτημα της, ε, δια, της διερεύνησης νέων λύσεων Υπάρχουν τέτοιου είδους ε, προβλέψει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε το εκπαιδευτικό σύστημα να στραφεί περισσότερο προς την ε, απασχόληση και τις θέσεις εργασίας. Και δεύτερον, για το μέλλον, γιατί ασφαλώς ε, τους επόμενους μήνες θα μπορέσετε να ορίσετε τα ορόσημά σας για το επόμενο διάστημα. Έχουμε κάνει τη συζήτηση για το πακέτο για τις τηλεπικοινωνίες και αυτό που διαπιστώνω εγώ είναι ότι υπάρχει και το πολιτιστικό ε, ενδιαφέρον από, την πλευρά του content, ε, από την πλευρά της βιομηχανίας παραγωγής πολιτιστικού υλικού που όμως μέσα στις προτάσεις δεν έχει λάβει επαρκή υποστήριξη και έμφαση. Σκοπεύετε λοιπόν εσείς να προβάλλετε περισσότερο αυτές τις, ε, αυτή τη διάσταση του πολιτιστικού περιεχομένου. Γιατί έχει σημασία, πέρασε πάρα πολύ γρήγορα μέσα από τις προτάσεις ε, πολύ βιαστικά δηλαδή μέσα από τις προτάσεις που έφτασαν στο Κοινοβούλιο και θα ήθελα να δοθεί περισσότερη έμφαση στο content, στο πολιτιστικό περιεχόμενο. Επίσης, πάλι στον χώρο των οπτικοακουστικών και με το βλέμμα προς, ε, το βλέμμα προς το μέλλον. Έχουμε αναλάβει δύο εκθέσεις όπου βρισκόμαστε τώρα σε μια φάση διαβούλευσης ε, για την πράσινη βιβλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το πολιτιστικό περιεχόμενο όπου θα πρέπει να ε, λυθούν διάφορες εμπλοκές που έχουμε στον τομέα αυτών. Και γι' αυτό θέλω να ρωτήσω πώς, τι είδους οδηγίες θα δώσετε για τη σχετική γενική διεύθυνση, πώς θα τηρεί, τι στάση θα τηρήσει δηλαδή, στον τομέα αυτών. Η κυρία Μακλάρκιν. Ευχαριστώ και ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία την τελευταία πενταετία και τις προσπάθειές σας να ε, πλαισιώσετε το έργο μας και την χρηματοδότηση που διαθέτουμε. Ελπίζουμε ότι αυτό θα φέρει αποτέλεσμα στα επόμενα χρόνια. Επίσης, ιδιαίτερα θέλω να υπογραμμίσω τη σημασία που αποδίδουμε εμείς ως Επιτροπή, της πιστεύω τουλάχιστον, στους νέους και τη φωνή των νέων που πρέπει να ακούγεται. Γι' αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε να δίνουμε τη σχετική έμφαση στη δουλειά μας όπως προχωράει. Χαίρομαι που παραμένει αυτή η υποστήριξη της διάστασης των νέων εγώ βλέπω ότι ωστόσο δεν υπάρχει επαρκή έμφαση στην επαγγελματική κατάρτιση. Πολλά λέμε για την ανώτατη εκπαίδευση, πολλά λέμε για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Πολλέ όμω θέσει εργασία θα πρέπει να βρούνε και μία θέση στην κοινωνία μα για του νέου. Και πρέπει να κοιτάξουμε περισσότερο του τρόπου να προαγάγουμε αυτή την επαγγελματική κατάρτιση, που σημαίνει και θέσει εργασία, που σημαίνει και νέε περισσότερε δεξιότητε για του νέου μα ώστε να μπορέσουν να μπουν στον επαγγελματικό βίο. Και θα ήθελα Επίσης να υπογραμμίσω τη σημασία του να συνδεθούν όλα αυτά με, την το ψηφιακό θεματολόγιο ώστε να φέρει αποτέλεσμα αυτό για τις κοινωνίες μας σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά πάνω απ' όλα για τους νέους. Εκπαίδευση, δυνατότητα επιχειρησιακής δραστηριότητας, ε, διαγραμμικής στο διαδίκτυο και ούτω καθεξής. Ξέρω ότι είναι γνωστή η θέση μου ότι δεν πρέπει να ενισχύονται τα κονδύλια στον προπολογισμό από τη θέση μου συντηρητική, αλλά πάνω απ' όλα πιστεύω ότι πρέπει να αξιοποιούνται τα εφιστάμενα κονδύλια κατά τρόπο σωστό και όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικό και βέβαια και για τον αθλητισμό θα πρέπει να δώσουμε έμφαση. Γι' αυτό θέλω να ρωτήσω πώς σκοπεύετε να αξιολογείτε, να κάνετε μια διαρκή ε, αξιολόγηση της αποδοτικότητας των κονδυλίων και των προγραμμάτων. Δηλαδή πρέπει, να και δεν έχουμε και τόσο πολλά κονδύλια, να βεβαιωνόμαστε ότι τα χρήματα τα οποία χρησιμοποιούμε αξιοποιούνται στο βέλτιστο δυνατό βαθμό, το επιθυμητό αποτέλεσμα και το καθεξής. Και νομίζω ότι η υποστήριξη της δημιουργικής ε, παραγωγής, της υποστήριξης ε, του κλάδου των, ε, των ταινιών και ούτω καθεξής παραγωγικής δηλαδή πνευματικής δραστηριότητας μπορούν να στηρίξουν και την οικονομία μας και τους νέους μας. Μπορούμε λοιπόν στο μέλλον να περιμένουμε περισσότερες τέτοιου είδους επενδύσεις που θα υποστηρίξουν την πνευματική παραγωγή και τους νέους μας. Ευχαριστώ. Μπακ, κυρία Πρόεδρε. Ε, θα μιλήσω ελληνικά. Ε, Gentlemen, you are behind Mrs. Pagliadelli. Είστε μετά την κυρία Παλιαδέλη, κύριε μου, διότι σηκώστε το χέρι σας μετά την κυρία Παλιαδέλη. Δεν τα έχω μπερδέψει, ξέρω πάρα πολύ καλά και αγαπητέ μου, ξέρετε πόσο σας αγαπώ και πόσο δίκαιη είμαι. I'm I, see your so I'm very suspicious. Please, Παλιαδέλη. κυρία Πάκ για τον κύριο Τάκουλα ή τον κύριο Λόκεγκαρτ ε, στη σειρά. Ε, καλημέρα σας κυρία Βασιλείου, ευχαριστούμε πολύ για αυτή την ε, έτσι, η συνοπτική παρουσίαση της δραστηριότητας ε, ε, του, της Γενικής Διεύθυνσης που, στην οποία προείσταστε και την πολύ καλή συνεργασία δεν θα επαναλάβω επένους για τον τρόπο με τον οποίο συνεργαστήκαμε οι δύο θεσμοί για να μην θεωρηθεί ότι μεροληπτό λόγω και της κοινή μας ε, καταγωγής. Ε, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω τις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε ως Επιτροπή Πολιτισμού για θέματα τα οποία για μένα έχουν γίνει πια έμονες ιδέε, Γνωρίζετε την αδυναμία μα να υποστηρίξουμε ω Ευρώπη και λόγω και της επικουρικότητα, την ε, διεύρυνση των ανθρωπιστικών σπουδών και κυρίω τη χρηματοδότησή σα. Κάναμε προσπάθειε με την κυρία Κώστα και στο πρόγραμμα Horizon και στο πρόγραμμα Creative Europe να περάσουμε το, την πολιτιστική κληρονομιά ως έναν από τους τομείς τους οποίους και η επιχειρηματικότητα και τα προγράμματα και η ανανέωση των ε, προγραμμάτων των, των, ε, των πανεπιστημιακών ε, σπουδών ε, μπορούν να υποστηριχτούν. θεωρώ ωστόσο ότι η αναγγελία σας για την, μια πρωτοβουλία που αφορά σε ένα πρόγραμμα ή ξέρω πρόγραμμα για την πολιτική κληρονομιά είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντική ως legacy για, το επόμενο, ε, για την επόμενη Ευρωβουλή και τα, ε, γιατί πραγματικά επεξεργαζόμενη την ε, δημιουργική Ευρώπη, το Erasmus και το Horizon είδα πουθενά δεν έχουμε μια συνολική πολιτική που να αφορά όχι μόνο στην προστασία και την ανάδειξη για λόγους τουριστικούς αλλά και την έρευνα τη βασική, τη χρηματοδότησή της επομένως αυτή τη διαπιστημονική έρευνα πρόκειται για να σκαθεί, πρόκειται για ειδικέ ε, άλλες εφαρμογές τεχνολογικές που αφορούν την επεξεργασία του ε, υλικού αυτής της πολιτιστικής κληρονομιάς. Θεωρώ λοιπόν ότι η Ευρώπη δικαιούται και οφείλει ένα τέτοιο, μια τέτοια πρωτοβουλία. Αν θα μπορούσατε να μου δώσετε κάποια πληροφορία περισσότερη στο πλαίσιο αυτής της, να μας δώσετε αυτής της παρουσίας που μας κάνετε. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα ο κύριος Τάκ.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 δεν ξέρω πώς διάβασες το πρόσωπό μου προηγουμένως ή το πρόσωπο του κυρίου Γιατί Εμείς δεν σκεφτήκαμε τίποτα από αυτά που είπες, μεταξύ μας μιλάγαμε. Εν πάση περιπτώσει, να επανέλθω τώρα σε αυτά τα οποία συζητούσαμε. Θα ήθελα και εγώ ξεκινώντας να ευχαριστήσω την κυρία Επίτροπο για μια συνεργασία πολυετή και ιδιαίτερα ικανοποιητική το Erasmus Plus ε, πράγματι ε, θα πρέπει να το χαρακτηρίσω τον θρίαμβο των δύο σιδηρών ε, κυριών που βρίσκονται στο Προεδρείο αυτή τη στιγμή. Και η αύξηση επίσης του προϋπολογισμού που μας αφορά είναι ένα τεράστιο επίτευγμα στη σημερινή συγκυρία. πράγματι πείσατε ότι αξίζει να επενδύει κανείς στην, στον πολιτισμό και στην εκπαίδευση στον δύσκολο αυτό καιρό τον οποίο ζούμε. Σας ευχαριστώ λοιπόν για μια ακόμη φορά. Και τα υπόλοιπα προγράμματα προωθήθηκαν με επιτυχία, αλλά το Erasmus Plus επιμένω ότι ήταν η κορονίδα της προσπάθειάς σας είναι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έλεγα το χαρτοφυλάκιό σας ένα ιδιαίτερα δύσκολο χαρτοφυλάκιο και γι' αυτό εγώ από την αρχή επέμεινα να πάρω μέρος σε αυτήν εδώ την Επιτροπή για να μπορέσω να πιέσω ε, η εκλογής μου και οι φίλοι μου στην Φιλανδία το θεώρησαν, την αιμονή μου αυτή την θεώρησαν λίγο περίεργη. Και κάποιοι πολιτικοί μου φίλοι σε εισαγωγικά είπαν ότι τελικά το Erasmus Plus ήταν το βασικό επίτευγμα της προηγούμενης αυτής πενταετούς περίοδου. Αυτοί που με ηρωνεύθηκαν σε μια κάποια πρώτη φάση τώρα πλέον αντιμετωπίζουν διαφορετικά την προσπάθειά μας τα τελευταία χρόνια. Δεν θα πρέπει να υποτιμηθεί ποτέ το βάρος και η σημασία της παιδείας και του πολιτισμού. Είναι ζωτική ανάγκη να συνεχιστεί η συνεργασία ανάμεσα στο Κοινοβούλιο και την Επιτροπή στον τομέα του πολιτισμού στρεφόμενος τώρα ε, μετά από αυτά τα λίγα λόγια ευχαριστίας στο μέλλον. Δεν ξέρω, ίσως μετά τις εκλογές να έχω τη χαρά να βρεθώ πάλι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ελπίζω να πείσω τους εκλογείς μου γι' αυτό. Και γι' αυτό θα ήθελα να ρωτήσω, να κάνω μια ερώτηση μπορείτε να μου πείτε τις τρεις βασικές προτεραιότητες τις οποίες θεωρείτε ότι πρέπει να επιδιώξουμε στον τομέα που σας αφορά στο επόμενο κοινοβούλιο, στην επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο. Ποια είναι τα τρία βασικά θέματα τα οποία θα θέλατε να επιδιώξουμε να προωθήσουμε αν ξαναείμαστε εδώ. Πανέρχομαι στο θέμα του αθλητισμού. Ε, ξέρετε ότι ο αθλητισμός παρουσιάζει ένα τεράστιο δυναμικό και στον τομέα της υγείας και στον τομέα της κοινωνίας. Ε, τι μπορούμε να κάνουμε για να πείσουμε τα κράτη-μέλη να δώσουν μεγαλύτερο βάρος και σε κοινοτικό επίπεδο στα του αθλητισμού. <clears throat> Λοιπόν, σας ευχαριστώ ε, Ντόρις και κυρίως Επίτροπε για τη συνεργασία τα τελευταία χρόνια. Σας ευχαριστώ και πάλι. Εύχομαι ό,τι καλύτερο στο μέλλον. Ευχαριστώ. Χάνω όποτε χρειαστώ να επισκεφθώ την Λαπωνία, ξέρω που θα σε βρω. Ο κύριος Λόκεγκαρτ. Thank you. Yet another elder member. Yes. Well, uh, Ευχαριστώ. Θα είμαι σύντομος γιατί τα περισσότερα που ήθελα να πω έχουν ήδη υποθεί. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την αξιότιμη κυρία Επιτροπό για την εξαιρετική της δουλειά, για την εξαιρετική συνεργασία με εμάς ε, και αυτό το οποίο θα πρέπει να τονίσουμε είναι το Erasmus ΣΥΝ. Αυτό είναι η τεράστια μεταρρύθμιση, το είπαν και οι προηγούμενοι ομιλητές. Είναι εξαιρετικά σημαντικό, μια τεράστια μεταρρύθμιση και νομίζω ότι όταν οι ιστορικοί αναλύσουν αυτή την πενταετή θητεία θα δουν ότι με ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα ήταν αυτό, το Erasmus σύν, ε, Το είπε και ο Χάνου και στη δική μου χώρα, στη Δανία. Είναι ένα από τα τρία βασικότερα ε, ζητήματα, ένα από τα τρία βασικότερα επιτεύγματα που γνωρίζει η κοινή γνώμη. Είναι ένα από τα τρία θετικά που αναφέρει ο κόσμος για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όποτε μιλήσει θετικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αραιά και που βέβαια. Τέλος πάντων. Από εκεί και πέρα, θα ήθελα να θέσω και ένα άλλο θέμα. Όπως και εσείς, να τονίσω τον ρόλο του πολιτισμού και της κουλτούρας ε, στην χάραξη της πολιτικής. Το σωστό ερώτημα που τίθεται είναι πώς θα το πετύχουμε αυτό. Ε, να περιλαμβούμε δηλαδή την κουλτούρα και τον πολιτισμό στις πολιτικές μας. Είναι καλή η δυναμική αυτή τη στιγμή και εσείς και όλη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πέτυχε. Ε, πέτυχε να θέσει την κουλτούρα σε, ε, ψηλά στον κατάλογο προτεραιοτήτων της πολιτικής ατζέντα. Ειδικότερα σήμερα σε καιρούς κρίσης. Άρα το ερώτημα που τίθεται είναι τι θα κάνουμε τα επόμενα πέντε χρόνια μετά την ανανέωση της κοινοβουλευτικής θητείας. Ήσασταν ε, παρούσα ε, πέρσι τον Απρίλιο όταν ξεκινήσαμε αυτό το project ε, για την χάρτα, την πολιτιστική για την Ευρώπη και μετά από δύο εβδομάδες στο Βερολίνο είχαμε το project Self Europe πριν από δύο εβδομάδες Βλέπετε δηλαδή ότι όσοι ασχολούνται με την κουλτούρα και τον πολιτισμό προσέχουν ιδιαίτερα τι κάνουμε. Ε, μπορούμε να τους προσεγγίσουμε. Τι θα κάνει λοιπόν η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα επόμενα πέντε χρόνια έτσι ώστε αυτές οι ιδέες να μεταφραστούν σε συγκεκριμένες πράξεις. Πώς θα προχωρήσουμε από εδώ και στο εξής που έχουμε όλες αυτές τις ιδέες, τις σκέψεις, τα προγράμματα πώς ο κόσμος του πολιτισμού θα καταφέρει ε, να κάνει τη φωνή του να ακουστεί ε, για συγκεκριμένα ζητήματα και μάλιστα σε τον ε, υψηλότερο πολιτικό επίπεδο. στις επίσημες δομές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι το ερώτημά μου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Νομίζω η κυρία Κώστα ήθελε το λόγο. Σας ευχαριστώ για την προσπάθεια που κάνατε κυρία Βασιλείου. Εγώ αναγνωρίζω μια τεράστια προσπάθεια και είδα ότι είχατε πραγματικά όραμα, ήσασταν διαθέσιμοι απέναντι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, απέναντι στις προτάσεις μας και σταθήκατε πάντα με επικοδομητικό τρόπο ακόμα και στις κριτικές τις οποίες σας έχουμε απευθύνει. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να σας ευχαριστήσουμε γι' αυτό. Ευχαριστώ επίσης και την κυρία Πάκα για το πάθος, την ε, προσπάθεια που έκανε και μια κάποια ηρωνία την οποία ε, μερικές φορές χρησιμοποίησε για να δουλέψουμε σωστά. Αυτό που πρέπει να υπογραμμίσει κανείς σε σχέση με τις προοπτικές και τα βήματα τα οποία έχουν γίνει και στον τομέα της παιδείας και στον πολιτισμό δεν είναι τίποτα δεδομένο, δεν πρέπει τίποτα να θεωρηθεί δεδομένο. Ε, πράγματι ο πολιτισμός βοηθάει στην ε, συνειδητοποίηση της ταυτότητας, στην ανάπτυξη, την οικονομική και στην καινοτομία. Αλλά ξέρουμε ότι έχουμε ζήσει κάποιες αντιφάσεις τα τελευταία χρόνια, αυτά τα οποία κάναμε εμείς εδώ στον τομέα της Creative Europe, και σε τομείς ε, στο επίπεδο πολιετούς προγραμματισμού, όπως μας είχε θυμίσει, μας θύμισε και η κυρία Παλιαδέλη. Σε άλλους τομείς τα πράγματα πήγαν με διαφορετικό τρόπο. Και γι' αυτό όμως με τη δική σας προσπάθεια το Horizon 2020 ενέταξε και θέματα που αφορούν την καινοτομία, που αφορούν ε, το, ε, την πολιτιστική κληρονομιά και ήταν μια καλή προσπάθεια και εκεί παρά τις δυσκολίες και ε, στην αρχή στον τομέα των διαφθορτικών ταμείων δεν υπήρχε καμία αναφορά στα θέματα του πολιτισμού. Παρ' αυτά βοηθήσαμε έτσι ώστε να ενταχθεί και ο πολιτισμός ε, εν μέρη τουλάχιστον στον τομέα αυτό. Έχει μεγάλη σημασία λοιπόν σε όλους τους τομείς και της οικονομικής ανάπτυξης και της έρευνας να μην χάνουμε το στόχο του πολιτισμού και η ανάπτυξη θα πρέπει να είναι ε, ένας, ε, μια ανάπτυξη ολοκληρωμένη που να λαμβάνει υπόψη και την πολιτιστική πραγματικότητα. Ο ρόλος του πολιτισμού λοιπόν είναι εγκάρσιος γενικά σε όλα αυτά τα θέματα και όχι μόνο κάθετος. Τώρα για το Creative Europe και επανέρχομαι σε αυτά τα οποία είπε η συνάδελφος κυρία Τρούπελ. Ένα σημαντικό θέμα στις επιλογές οι οποίες γίνονται στις διάφορες χώρες έχει σημασία σε επίπεδο του desk της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να υπάρξει μια διαθεσιμότητα επικοινωνίας με διαφορετικούς κάθε φορά ομιλητές γιατί είναι διαφορετικές οι κατανομές των αρμοδιοτήτων σε κάθε χώρα και αυτό έχει σημασία να μην αποκλείσουμε κανένα. Τώρα, ε, να επανέλθω στο θέμα των δικτών. Για τους δίκτες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει κάποιους δείκτες για τον τομέα του πολιτισμού και της δημιουργικότητας. Είναι αρκετά σημαντικό αυτό, γιατί ναι μεν αυτό στον τομέα τον ραδιοτηλεοπτικό ας πούμε είναι σχετικά προχωρημένο, στον υπόλοιπο τομέα, στον πολιτιστικό τομέα δεν έχουμε αυτούς τους δείκτες σωστά διαμορφωμένους. Τώρα για την πρωτοβουλία, για την πολιτιστική κληρονομιά. Η Ιταλική Προεδρία θέλει να δώσει μεγάλο βάρος ε, στην προσπάθεια αυτή και χαίρομαι που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα είναι διαθέσιμη. Merci, Madame la Présidente. Κυρία τελευταία ομιλήτρια, πολλά υπόθηκαν από τους συναδέλφους και δεν θα ήθελα να τα επαναλάβω να σταθώ σε ένα θέμα που θεωρώ σημαντικό και αφορά δύο επίτροπες, όχι μόνο τη δική μας, είναι το θέμα της νεότητας. Ε, βρισκόμαστε σε ένα σταυροδρόμι. Ξέρουμε ότι αμφισβητείται το ευρωπαϊκό όραμα, υπάρχει μια απομάκρυνση και αδιαφορία του κόσμου και των νέων. Ε, οι νέοι μου λένε σήμερα ότι τι είναι η Ευρώπη, δεν πιστεύουμε πια στην Ευρώπη. Για το θέμα λοιπόν της νεότητας υπάρχει κάτι το πάρα πολύ σημαντικό, είναι το Ταμείο Εγγύησης για, την, για τους νέους, έτσι ώστε τα κράτη-μέλη να επιτρέψουν στους νέους μετά από την εκπαίδευσή τους να βρουν μια λύση στον τομέα της απασχόλησης. Θα ήθελα εδώ να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε εμείς στον τομέα του πολιτισμού, στον τομέα των μέσων ενημέρωσης και της εκπαίδευσης. Πώς μπορούμε έτσι ώστε να εκμεταλλευτούμε το μέσο αυτό έτσι ώστε αυτή η εγγύηση να μην παραμείνει ένα ουτοπικό πρόγραμμα, αλλά να γίνει πραγματικότητα και στους τομείς μας, στους τομείς που μας ενδιαφέρουν και να μην αγνοηθεί ε, η οικονομική πραγματικότητα της εκπαίδευσης και του πολιτισμού. Και εγώ έχω μία μικρή ερώτηση, λέει η Πρόεδρος. Και μάλιστα πολύ πρακτική ερώτηση. Έχουμε σημειώσει ότι δεν θέλουμε να προάγουμε ετήσιες εκδηλώσεις. Υπάρχει κάτι το διετές, είναι διετής εκδήλωση κάθε δύο χρόνια φερπίνει οι Special Olympics που εμένα με ενδιαφέρουν πάρα πολύ. Όχι οι Para Olympics, οι Special Olympics που κατά τα άλλα δεν έχουν υποστήριξη. Είναι αναδιαιτία. Αυτή η απαγόρευση λοιπόν της ε, υποστήριξης ε, ετησίων ε, ενιαυσίων ή μάλλον ετησίως επαναλαμβωμένων εκδηλώσεων ισχύει ή θα μου πείτε όπως ο Πάπας άλλο ετήσιος και άλλος διετής. Αυτή είναι η δική μου ερώτηση. Έχετε και τι υπόλοιπε Ανδρούλα, το λόγο. Με μεγάλη χαρά άκουσα ότι πάρα πολλοί από εσά έθεσαν το ερώτημα ε, της ανεργίας των νέων. Και βέβαια αυτή είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Και σας διαβεβαιώ ότι και εγώ προσωπικά και ο Επίτροπος Άντορ και ο Πρόεδρος Μπαρόζο θεωρούμε ότι αυτή είναι η κύρια ε, προτεραιότητά μας. Πώς θα αντιμετωπίσουμε την τεράστια πρόκληση της ανεργίας των νέων. Και βέβαια η εγγύηση για τους νέους είναι ένα πολύ καλό εργαλείο. Ένα μέσο έτσι ώστε οι νέοι είτε να βρουν δουλειά, είτε να συνεχίσουν τις σπουδές τους, είτε να βρουν ε, ε, θέση για κατάρτιση, για μαθητεία, για άσκηση και ζητήσαμε από όλα τα κράτη-μέλη μέχρι τα τέλη της περασμένης χρονιάς να υποβάλουν τα σχέδιά τους για τον τρόπο τον οποίο θα εφαρμόσουν αυτό το πρόγραμμα για την εγγύηση των νέων. Και το έκαναν. Τα σχέδια αυτά τα έχουν ελέγξει λοιπόν οι υπηρεσίες μας και προσπαθούμε να ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη αυτή τη στιγμή για να τα υλοποιήσουν, να τα εφαρμόσουν αυτά τα σχέδια. Και έχουμε και τα 6 δις ευρώ με τα οποία έχει πρικιστεί ο προϋπολογισμός για τα επόμενα χρόνια στο πλαίσιο του ε, πολιετούς ε, δημοσιονομικού ε, σχεδιασμού. Και τα κράτη-μέλη που δικαιούνται αυτά τα χρήματα για να εφαρμόσουν την εγγύηση για τους νέους θα τα πάρουν την πρώτη και την δεύτερη χρονιά αυτά τα χρήματα. Το 2014 και το 2015 θα λάβουν αυτά που δικαιούνται για να εφαρμόσουν αυτό το πρόγραμμα. Δεν είναι όμως μόνο ε, το πρόγραμμα αυτό που έχει σημασία. Δεν τελειώνει εκεί το πράγμα. Όπως είπα και προηγουμένως, έχουμε ξεκινήσει και τη συμμαχία για την μαθητεία, για την άσκηση. Γιατί πολύ συχνά, ξέρετε, οι νέοι που είναι άνεργοι υστερούν από πλευράς προσόντων. Πρέπει να τους φρικίσουμε με προσόντα, με εργασιακή εμπειρία για να μπορούν να βρουν θέση απασχόλησης. Όλα αυτά συνδέονται μεταξύ τους και είναι και άρρηκτα συνδεδεμένα με τις προσπάθειές μας για το διτό σύστημα εκπαίδευσης το οποίο σαφέστατα έχει αποδειχθεί ως ένα πολύ επιτυχημένο σύστημα. Προσπαθούμε να ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη από τις ε, χώρες ε, της Ευρώπης του Νότου που δεν είχαν μεγάλη παράδοση επαγγελματικής κατάρτισης ε, στο εσωτερικό τους να συνάψουν εταιρικέ σχέσεις με άλλες χώρες όπως η Γερμανία, η Αυστρία, η Δανία που έχουν μακρά παράδοση στην εκπαιδευτική και επαγγελματική κατάρτιση έτσι ώστε να μάθει ο ένας από των άλλων. Και ενθαρρύνουμε τις χώρες του Νότου να αξιοποιήσουν ε, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για να ενισχύσουν τα εθνικά τους συστήματα για την επαγγελματική κατάρτιση. Ενθαρρύνουμε τις επιχειρήσεις επίσης να αναλάβουν δέσμευση. Δέσμευση να δημιουργήσουν προγράμματα μαθητείας και άσκησης και πιο πολυάριθμα και πιο ποιοτικά. Και Αυτά είναι νέα στοιχεία γιατί τώρα οι εμπλεκόμενοι φορείς για πρώτη φορά συνεργάζονται στενά, δουλεύουν μαζί για να έχουμε περισσότερες δυνατότητες μαθητείας, άσκησης, ε, όχι μόνο περισσότερες αλλά και πιο ποιοτικέ μέσα στο εσωτερικό, στους κόλπους των επιχειρήσεων. Και αυτό θα βοηθήσει, όλα αυτά θα βοηθήσουν πολύ ε, τους νέους. Βεβαίως το εκπαιδευτικό σύστημα έχει ένα τεράστιο ρόλο που καλείται να διαδραματίσει για να δώσει στους νέους τις εμπειρίες, τα προσόντα, τις δεξιότητες που χρειάζονται όχι μόνο για να βρουν θέση απασχόλησης αλλά ε, και που χρειάζονται για όλη την υπόλοιπη τους ζωή. Και μιλούμε για όλα ε, για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Έχουμε μια πρωτοβουλία για πολύ ε, από νωρίς ένταξη στο σχολικό ε, σύστημα και στην φροντίδα. Δηλαδή ένταξη στην ε, θεσμοθετημένη προσχολική φίτηση αν θέλετε. Γιατί πολύ, από πολύ νωρίς τίθενται τα σωστά θεμέλια, σωστές βάσεις. Και έχουμε πολύ μεγάλο συσχετισμό δείχνουν οι έρευνες μεταξύ των επιδόσεων των παιδιών και της προσχολικής αγωγής. Δηλαδή, όσοι έχουν φοιτήσει σε δομές προσχολικής αγωγής για πάνω από ένα χρόνο, έχουν στη συνέχεια καλύτερες επιδόσεις στην σχολική εκπαίδευση αυτή αυτή και έχει αποδειχθεί ε, σαφέστατα ο συσχετισμός μεταξύ των δύο. Τώρα, ως προς το πολιτιστικό περιεχόμενο. Όντω, οι νέε τεχνολογίε δεν πρέπει να υπονομεύουν τι αρχέ μα. Αυτό είναι το βασικό. Λέμε δηλαδή ότι κάθε δημιουργό πρέπει να αμείβεται για την δημιουργία του. Διότι δεν μπορεί κανείς να βασίζεται στις ψηφιακές τεχνολογίες χωρίς να έχει ε, ποιοτικό περιεχόμενο μέσα σε αυτές. Και γι' αυτό συνεργαζόμαστε στενά με τον Επίτροπο κύριο Μπαρνιέ και την Επίτροπο κυρία Νέλη Κρούς για να ε, βρούμε σωστά ισορροπημένες λύσεις. Εγώ θέλω να διατηρήσουμε αυτή την αρχή που ε, μας χαρακτηρίζει από πλευρά δημιουργών. Οι δύο άλλοι επίτροποι ασχολούνται με διαφορετικά θέματα και γι' αυτό θέλουμε να βρούμε τη χρυσή τομή. Και σας παραπέμπω στο εξής ε, το Licenses for Europe, οι άδειε για την Ευρώπη, είναι ένα πολύ καλό εργαλείο για να το πετύχουμε αυτό που θέλουμε, αυτό το σημείο ισορροπία. Έχουμε συνεργαστεί οι τρει επίτροποι για την ψηφιακή ατζέντα, για το πολιτιστικό περιεχόμενο και καταλήξαμε σε πολύ συγκεκριμένα αποτελέσματα. Δεν είναι βέβαια και ε, τέλεια η έκβαση των διαπραγματεύσεων και των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων, σαφέστατα. Όμω υπάρχουν αποτελέσματα. Όταν υπάρχει στενή συνεργασία, αυτό έχει φανεί ξεκάθαρα, μπορούμε να έχουμε ψηφιακή τεχνολογία, ναι, αλλά ε, και ε, προστασία των ευρωπαϊκών αξιών ε, τις οποίες στερνιζόμαστε. Τα προγράμματά μας αξιολογούνται συνεχώς. Δεν μπορούμε να πούμε ότι το όποιο πρόγραμμα, είτε το Erasmus Συν, είτε το Δημιουργική Ευρώπη, ε, το φτιάχνουμε, το συντάσσουμε, το χαράσουμε και τέλος. Όχι. Ε, τα παρακολουθούμε και διασφαλίζουμε ότι γίνεται σωστή η εφαρμογή τους. Ε, γίνεται αξιολόγηση και εσωτερική από εμάς αλλά και από εξωτερικούς αξιολογητές για να δούμε την αξία αυτών των προγραμμάτων, των έργων, των σχεδίων. Πριν την υιοθέτηση των νέων προγραμμάτων είχαμε εξωτερική αξιολόγηση σε μεγάλο βάθος για να δούμε τι δουλεύει και τι δεν δουλεύει, τι λειτουργεί και τι δεν λειτουργεί και γι' αυτό κάναμε streamlining στις δράσεις που προτείναμε βάσει των νέων προγραμμάτων για να μπορέσουμε να κάνουμε και σωστή αξιολόγηση. Η επένδυση στην εκπαίδευση. Επιτρέψτε μου να σας υπενθυμίσω ότι στις συστάσεις ανακράτος που υιοθετούμε κάθε χρόνο η Επιτροπή και μετά περνάνε στο Συμβούλιο δεν παραλείπουμε να διατυπώσουμε συστάσεις για επενδύσεις στην εκπαίδευση. Διότι και σε περίοδους κρίσης ακόμη θα πρέπει να επενδύουμε στην, στην εκπαίδευση. Αλλά πιο σημαντικό απ' όλα να επενδύουμε με τρόπο ευθύ. Διότι πολύ συχνά πολλές χώρες επενδύουν πολλά στην εκπαίδευση αλλά με πολύ συχνά αποτελέσματα. Γι' αυτό θα πρέπει και να ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη να μην ε, περικόπτουν τους προπολογισμού τους για την ε, εκπαίδευση, αλλά ταυτόχρονα να ε, εστιάζουν το ενδιαφέρον τους στα σημεία που διαπιστώνονται και οι αδυναμίες. Και γι' αυτό από τα 28 τα 18 κράτη-μέλη, από ό,τι θυμάμαι την προηγούμενη φορά, είχαν λάβει σοβαρές συστάσεις για την εκπαίδευση. Και γι' αυτό υπογραμμίζω ότι η εκπαίδευση είναι κεντρική σημασία ε, θέμα για την χάραξη πολιτικής. Ο κύριος Στάκουλα με ρώτησε τι προτεραιότητες έχω για την προσεχή επιτροπή στον χώρο του πολιτισμού. Πολλές προτάσεις θα είχα, αλλά θα ξεκινούσα με την πολιτιστική κληρονομιά. Το είπα ήδη και με ενθαρρύνει και η κυρία Παλιαδέλα να το επαναλάβω, ότι η πολιτιστική κληρονομιά από την εμπειρία που έχω τα τελευταία 4-5 χρόνια, Καταλήγω στο συμπέρασμα ότι είναι πολύ σημαντική η πολιτιστική πληρονομιά και επιτρέπει στους πολίτες να την εκτιμούν και να βλέπουν πόσο μεγάλη συμβολή έχει στην ανάπτυξη των πόλεων, των περιφερειών, των χωρών η προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς έχει πολύ μεγάλη σημασία λοιπόν και γι' αυτό αποφασίζω πριν από το τέλος της θητείας μου να προβώ σε μια ανακοίνωση για την πολιτιστική κληρονομιά προκειμένου να ενθαρρύνω την ανάπτυξη σοβαρών συζητήσεων κράτη-μέλη και εμπλεκόμενοι φορείς ώστε να δούμε πώς μπορούμε περισσότερο να προσδώσουμε αξία σε μια Ευρώπη της ενότητας και της ε, ποικιλία ενωμένη στη διαφορά. Και βέβαια το δεύτερο θέμα είναι το πώς μπορούμε να πείσουμε με επιχειρήματα ότι μπορούν να φέρουν καλά αποτελέσματα ο πολιτισμός και η εκπαίδευση στην Ευρώπη. Το συζητούμε βέβαια πολύ συχνά, αλλά το κάθε κράτος μέλος με διαφορετικό τρόπο προσμετρά την, ε, τον αντίκτυπο του πολιτισμού. Ξεκινάμε λοιπόν με τη Eurostat καταρχάς να διατυπώσουμε κοινού ορισμούς για το τι εννοούμε πολιτιστική και δημιουργική βιομηχανία ή κλάδος, ώστε να ξέρουμε ότι μιλάμε για το ίδιο πράγμα όταν συζητούμε. Και δεύτερον, όπως είπα και νωρίτερα, ξεκινούμε μια διαρκή αναζήτηση με το κοινό κέντρο ερευνών, μια διαρκή έρευνα, ώστε να προσφέρουμε στα κράτη-μέλη τα πορίσματα των ερευνών αυτών. Και τρίτον, θα ήθελα η ευρωπαϊκή παραγωγή ταινιών να υπερκεράσει την αμερικανική τη αυτή. Βεβαίως έχουμε υποστηρίξει πάρα πολύ την παραγωγή ταινιών στην Ευρώπη, παρόλα αυτά όμως ε, ακόμα πολύ. Και ιδιαίτερα εμένα με ενδιαφέρει πολύ το θέμα της ε, γνώσης, της χρήσης των ε, μέσων μαζικής ενημέρωσης και της γνώσης σχετικά με τις ταινίε. Είχα συμμετάσχει σε μια μεγάλη διάσκεψη στο Άμστερνταμ για το θέμα αυτό και με μεγάλη χαρά είδα τα μεγάλα προγράμματα και σημαντικά προγράμματα που αναπτύσσονται στον τομέα αυτών. Μίλησα λοιπόν με τον πρόεδρο του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της Ελλάδας και στο προσεχέ Συμβούλιο, ε, Συμβουλίου Παιδείας, με την Προεδρία της Ελλάδας, ο οποίος ε, συμφώνησε στην επόμενη συνεδρίαση να προσκαλέσει εκείνους οι οποίοι έχουν λάβει τη σχετική πρωτοβουλία στο Ηνωμένο Βασίλειο με ένα πιλωτικό, πιλωτικό πρόγραμμα ε, στη συνεργασία με 27 σχολεία, ενημέρωση, γνώση για την ε, κινηματογραφική παράδοση και τώρα έχουν αναπτύξει μια ε, εκδήλωση που έχει φτάσει κάθε εβδομάδα να καλύπτει πάνω από 30.000 σχολεία στο Ηνωμένο Βασίλειο. Να μια καλή ευκαιρία λοιπόν για βέλτιστες πρακτικές που κοινοποιούνται και ενθαρρύνεται να αξιοποιούνται και σε άλλα κράτη και η Γερμανία επίσης. Ο Βιμ ξέρουμε ότι ενδιαφέρεται ιδιαίτερο για το θέμα αυτό. Θέλουμε να το προαγάγουμε, να προαγάγουμε αυτή την ε, προσέγγιση στον κινηματογράφο. Γιατί αν μπορέσουμε από νωρί να δείξουμε στους νέους μας τον τρόπο να αξιολογούν την ποιότητα και τις αξίες της, ελληνικής, της ευρωπαϊκής κινηματογραφικής παραγωγής, μπορούμε να επιτύχουμε πάρα πολλά. Για τον κύριο Λόκερκαρτ. και εσείς και εγώ και η Ντόρις έχουμε εργαστεί σκληρά για να διατυπώσουμε ένα νέο λόγο για την Ευρώπη και αυτό πρέπει να το συνεχίσουμε. Δεν αρκεί να κάνουμε 5-6 εκδηλώσεις στην Ευρώπη. Πρέπει τακτικά να έχουμε ε, την ε, οργάνωση τέτοιου είδου εκδηλώσεων και εγώ που πηγαίνω ενθαρρύνω τους συνομιλητές να οργανώνουν τέτοιου είδου εκδηλώσεις γιατί δεν είναι απαραίτητο να έρθει πάντα η μεγάλη γνωστή προσωπικότητα ή ο αρχηγός κυβέρνησης να μιλήσει και να συμμετάσχει στην εκδήλωση. Όμως ο διάλογος, η επαφή, η επικοινωνία και η συνομιλία με τον πολίτη έχει πολύ μεγάλη σημασία. Και θα ήθελα επίσης να ενθαρρύνω και τους ε, καλλιτέχνες, τους ανθρώπους του πνεύματος και της διανόησης να υψώνουν πιο συχνά τη φωνή. Φαίνεται ε, να περιορίζεται στο να εκδηλώνουν τις ε, θέσεις τους μόνο όταν διαπιστώνουν προβλήματα και ξέρουμε όταν προσπαθήσαμε παραδείγματι να εξασφαλίσουμε την πολιτιστική εξέρεξη από την TTIP στη συμφωνία με τις ε, ΗΠΑ. Ε, ξέρουμε τι είδους στάσεις ε, τηρούν όταν βλέπουν ότι δεν περιλαμβάνονται προγράμματα για τα μέσα. Αλλά δεν τους ακούμε πέραν της αντίδρασής τους να μιλούν θετικά για το πώς βλέπουν το θετικό ρόλο της, της πολιτιστικής ταυτότητας της Ευρώπης, για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, για το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Αυτό πρέπει να αναζητήσουμε και πιστεύω ότι σε όλη την Ευρώπη μπορούμε και πρέπει να πείσουμε τους ανθρώπους του πνεύματος και της διανόησης να μιλήσουν περισσότερο στο θέματα αυτά. Η δική μου ερώτηση για τις αιτήσεις, αιτήσεις επαναλαμβανόμενες αθλητικές εκδηλώσεις. Όχι, δεν αποκλείονται τελείως αυτές. Από αυτά που θυμάμαι τουλάχιστον είχαμε πει ότι γιατί ήδη μιλάμε με κάποιους αλλά θα πρόκειται για αγώνες. Δεν θα δίνουμε δηλαδή εμείς μια χορηγία ή μια δωρεά γιατί μας αρέσει μια εκδήλωση. Θα γίνεται, διορθώνει διαγωνισμός και οποιοδήποτε τελικά κερδίσει από τις ε, εκδηλώσεις ή τα, ε, τους αγώνες αυτούς, ε, τους αθλητικούς, θα λαμβάνει την χορηγία. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος, κύριε Επίτροπε. Θα προσθέσω και εγώ δύο λόγια, γιατί στρέφουμε το βλέμμα προς το μέλλον και θα μιλήσω γερμανικά. Πολλοί συνάδελφοι νομίζω δεν γνωρίζουν καν ότι διαθέτουμε μια νέα γενική διεύθυνση για την έρευνα Γενική Διεύθυνση Υπηρεσία Ερευνών, η οποία επαληθεύει όλα τα προγράμματα για να αναζητήσει την προσθέμενη τους αξία, την ευρωπαϊκή προσθέμενη αξία και η τελευταία που είδα εγώ, γιατί δεν έχει και πολύ καιρό που λειτουργεί, ήταν αυτή η οποία εξέταζε τον, το κόστος της απουσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε διάφορους τομείς, the cost σε διάφορους τομείς λοιπόν και νομίζω ότι εάν μαζί εργαστούμε για να κοιτάξουμε και αυτά τα οποία μας προσφέρουν οι συνάδελφοι αυτής της Γενικής Διεύθυνσης για την έρευνα, γιατί υπάρχουν πολλές δυνατότητες να βρούμε πού μπορούμε καλύτερα να δραστηριοποιηθούμε, τι είδους καλύτερο, καλύτερη αξία, περισσότερη αξία μπορούμε εμείς να προσφέρουμε. Υπάρχουν δυνατότητες. Αυτό ήθελα να σας ε, καταστήσω γνωστό. Και δεύτερον, Ξέχασα νωρίτερα να πω ότι η Επιτροπή κάνει πράγματα στα οποία δεν συμμετέχουμε, δεν θα έπρεπε μάλλον κανονικά να συμμετέχουμε, αλλά μας ε, καλεί. Επί παραδείγματι το βραβείο λογοτεχνίας, το Ευρωπαϊκό Βραβείο Λογοτεχνίας που είναι μια υπέροχη ιστορία, πολύ καλή. 12 με 13 κράτη αναέτος καλούνται να επιλέξουν έναν υποψήφιο και εδώ στα θέατρα, στα όμορφα μικρά θέατρα που έχουμε, γίνεται η απονομή των βραβείων. Και η Επίτροπος πάντοτε είχε την καλοσύνη να καλεί και την Επιτροπή μας, είτε με δική μου παρουσία, και με τον άλλων συναδέλφων, για να συμμετέχουμε. Ξέρουμε ότι υπάρχουν περιπτώσεις και εκδηλώσεις, οι οποίες δεν έχει προσκληθεί ποτέ το Κοινοβούλιο και γι' αυτό θέλω να σημειώσω ότι εσείς είχατε μια τελείως διαφορετική στάση και να υπογραμμίσω ότι πάντοτε μας προσκαλούσατε. Θα ήθελα επίσης να εκφράσω υποστήριξη για τα πολλά φεστιβάλ που έχουμε στην Ευρώπη και να πω ότι είναι μια πολύ καλή ιδέα να τα στηρίζουμε. Θα παρακαλούσα πάντως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο μέλλον να στρέψει το βλέμμα και προς τα θέατρα, τη θεατρική παραγωγή, όχι μόνο τα φεστιβάλ και ίσως θα ήταν καλό να δώσουμε περισσότερη έμφαση και σε αυτό. Τα φεστιβάλ ναι, τη λογοτεχνία ναι, αλλά μην αφήνουμε και το θέατρο στο περιθώριο. Πολλοί άνθρωποι του θεάτρου μου λένε συχνά «Μα δεν σας βλέπουμε ποτέ, δεν είσαστε ποτέ παρόντες». Είναι κρίμα αυτό νομίζω και ίσως μπορεί το προσωπικό σας, που σε τελευταία ανάλυση θα μείνει έστω και αν εσείς ενδεχομένως δεν επιστρέψετε, ε, να ασχοληθούν και με το θέμα αυτό και να το κοιτάξουν πιο προσεκτικά. Ένα άλλο που ήθελα επίσης να τονίσω, που είπε ο κύριος Λόκεγκαρτ, ήταν ότι ναι, είχαμε μια καλή εκδήλωση που μπόρεσε να φέρει κοντά ε, ανθρώπους της διανόησης του πνεύματος, επικεφαλής κυβερνήσεων, με τον κύριο Μπαρόσο, ακόμη παρόντα, πολύ καλά και πολύ χρήσιμη εκδήλωση και σημαντική. Αλλά πρέπει να συνεχίσουμε τέτοιου είδους ιδέες, γιατί υπάρχουν πολλές ιδέες που μπορούν να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο της ε, δουλειάς μας και νομίζω ότι ε, αυτή η ιδέα του Soul for Europe είναι μια ιδέα που μπορούμε να αξιοποιήσουμε. Και Ανδρούλα, το θίξαμε και νωρίτερα πόσο σημαντική είναι η κινηματογραφική παραγωγή. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το έχει αναγνωρίσει με το βραβείο Lux όπου οι συνάδελφοί μου μπορούν όλοι να πάνε και στα σχολεία και να το προβάλλουν σαν ένα απτό εργαλείο και παράδειγμα για το τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, να δείξουν την ταινία, να συζητήσουν ενδεχομένως το θέμα αυτό και να δώσουν και παραπάνω έναυσμα για μελέτη και αναλογισμό. Ε, θα ρηπίνει εκείνη η ταινία με τους ε, ε, τούντε στο άσυλο, στον Ντόβερ, ή η ταινία Φρέμντε που ήταν η σχετική με τους φόνους για λόγους τιμής. Συνεργασία λοιπόν με το κανάλι Άρτε, το βραβείο Λουξ, video on demand το οποίο διαθέτει για τρεις μήνες ε, στο διαδίκτυο την ταινία ή δυνατότητα για τα σχολεία και αυτή όλη η δυνατότητα για την επικοινωνία με τους πολίτες που δεν πρέπει να υποτιμούμε. Εδώ νομίζω μπορούμε και περισσότερο στα κράτη, στις πρωτεύουσες των κρατών μελών να δώσουμε έμφαση. Μεγάλη σημασία φυσικά έχει ο υποτιτλισμός. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να προβάλλουμε. Ακριβώς σε αυτό έχει κάνει το Άρτε πολύ μεγάλη δουλειά γιατί ανέλαβε το σχετικό ε, έργο. Τα τελευταία πέντε χρόνια λοιπόν έχουμε εργαστεί εδώ οι συνάδελφοι μαζί και θέλω να ελπίζω ότι οι συνάδελφοι που θα μείνουν και στην επόμενη θετία στην Επιτροπή μας θα συνεχίσουν τη δουλειά που έχουμε ξεκινήσει και εσάς, οι δικοί σας, ε, οι συνεργάτες, αγαπητή κυρία Επίτροπη, Επίτροπε, θα συνεχίσουν αυτή την κοινή προσπάθεια. Ευχαριστώ εδώ τους συναδέλφους ε, που έχουν ε, μπορέσει να έρθουν σήμερα. Ευχαριστώ εσάς θερμά, όπως και όλο σας το προσωπικό και επιτελείο, για την πολύ καλή συνεργασία σε όλους τους θεομείς, για την κατανόηση που επιδείξατε απέναντί μας πολλές φορές ίσως μερικές φορές ήμασταν, πώς το λέμε στα αγγλικά, rude, αγενείς. Χωρίς να θέλω όμως να είμαι προσβλητική. Ε, νομίζω ότι έχετε πια συνηθίσει πως ε, αυτά που σκέφτομαι τα λέω χήμα και εν πάση περιπτώσει, αλλά αυτό ίσως καμιά φορά χαλαρώνει και το κλίμα τρόπον την να. Ε, να, μερικές φορές μου λένε και διερμηνείς ότι μαζί μου περνάνε ωραία στην καμπίνα γιατί μπορούν και να διασκεδάσουν λίγο, να γελάσουν. Πάντως όπως και να είναι νομίζω ότι έχουμε περάσει μια πολύ καλή περίοδο μαζί, μια ε, περίοδο 4-5 ετών. Εύχομαι κάθε καλό και σε εσά προσωπικά για την περίοδο μετά την ολοκλήρωση των καθηκόντων σας ο Επιτρόπου. Ήταν πολύ καλή αυτή η δεύτερη θητεία, καλύτερη από την πρώτη που είχατε την υγεία, ο πολιτισμός νομίζω, η εκπαίδευση, η ψυχή της Ευρώπης. Ήταν αυτό το οποίο πραγματικά και σε εσάς ταιριάζει πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση. Ε, Περνάω γρήγορα στα διάφορα. Τίποτα. Κύριε Στάκουλα. Έλα, χάνω. Αγαπητοί φίλοι. Νομίζω ότι θα συμφωνήσουν όλοι μαζί μου. Θα τα ξαναπείς, λέει η Ντόρις. Είναι η σωστή μέρα σήμερα, 18 Μαρτίου. Χρόνια πολλά λοιπόν για τα γενέθλιά σου. Doris. Happy birthday to you. Thank you very much.